Νομίζω ότι μπορώ σήμερα να καλωσορίσω έναν έναν ονομαστικά τους παρόντες. Γιουπτσέβα, Χάουκ, Κάρενμπαχ, Σλίτερ, Γκερμπράντι, Γένζεν, τόσο ευάγριθμοι είμαστε. Α, και ο κύριος Σιμαντσκι, καλώς ήρθατε. Η σημερινή ημερήσια διάταξη δεν προβλέπει μεγάλες ψηφοφορίε τις έχουμε τη Δευτέρα. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε κάποια σημεία να επεξεργαστούμε σήμερα. Ρωτώ πρώτον λοιπόν για την έγκριση. Παρατηρήσεις ή προτάσεις για τροποποίηση. Όχι. Διερμηνία. Ο συνήθως πλην της εσθονικής και της μαλτεζικής. Συνεχίζω με τους τριμερείς διαλόγους. Έχουμε στις 4 Μαρτίου την οδηγία για το μέλι, όπου συμφωνήσαμε και έτσι 19 Μαΐου, Μαρτίου ψηφίζουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για να πάει στη δεύτερη σύνοδο του Απριλίου η ψηφοφορία. Έχουμε συμφωνία ως προς το σύστημα ανταλλαγής εκπομπών για τα αεροσκάφη. Στις 4 Μαρτίου επετεύχθη η συμφωνία. Δεν είναι σαφές ωστόσο αν θα την ακολουθήσουν όλες οι πολιτικές ομάδες. Το συμβαστικό κείμενο θα πρέπει να εγκριθεί εδώ στην Επιτροπή μας. Δεν όμως αφήσει ακόμα η κατάσταση. Παραμένει η ένταση της αναμονής. Μετά έχουμε το θέμα των λιμένων τον τριμερή διάλογο που εχθές επετεύχθη συμφωνία και εχθές ακόμη σε ένα θέμα που έχω την έκθεση την ΣΥΤΕΣ όπου διέκοψα για τρία λεπτά τον τριμερή διάλογο για να πω στο Συμβούλιο ότι είναι απαράδεκτο να διαγράφονται όλες οι κατεξουσιοδότης συμπράξεις και να αφαιρούνται όλες οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες του Κοινοβουλίου. Είπα ότι δεν πρόκειται να το δεχθούμε αυτό και ελπίζω να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα άλλες επιτροπές διακόπτοντας την συνεδρίαση. Όταν έχουμε σαφή εντολή για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χειριζόμαστε τα θέματα από εδώ και μπρο, πρέπει να το κάνουμε. Στο ΣΥΤΕΣ λοιπόν δεν χάσαμε τίποτα, δεν έχουμε πίεση χρονική και δεν δεχόμαστε να μας ε, αφαιρούν με τον τρόπο αυτό τα δικαιώματά μας. Μέσα σε τρία-τέσσερα λεπτά λοιπόν είχε κλείσει το θέμα. Και συνεχίζω πρακτικά της 27 28 η 22ης-23ης Ιανουαρίου. 23 παρατηρήσεις εδώ, όχι, εγκρίνονται. Και έτσι περνώ στο σημείο 4 για μια ανταλλαγή απόψεων που προβλέπεται σήμερα με το ελεγκτικό συνέδριο και τον κύριο Ιαν Κίνστ. Εφαρμογή του LIFE. Έχουμε την μόνιμη εισηγήτρια παρούσα εδώ. Πρέπει να πω ότι εγώ είμαι φαν του LIFE. Είναι ένα από τα μεγάλα, τις μεγάλες επιτυχίες της ε, πολιτικής μας. Είναι ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ανυπομονησία την ανάλυση σας και τις προτάσεις σας, τις συμβουλές που μπορεί να μας δώσετε. Ο Γιάννη Κίνης λοιπόν έχει τον λόγο πρώτος για να ακολουθήσει η Ιούτα Χάουκ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Yeah, thank you, Mr. Chairman. Thank you very much for the Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτή τη συνεδρίαση και να σας παρουσιάσω τα πορίσματα της έκθεσης περιθμών 15 για το 2013 που αφορά την συνιστόσα του περιβάλλοντος στο πρόγραμμα LIFE. Όπως θα ξέρετε, η ουσία των δαπάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον αφορούν πολλές πολιτικές. Το πρόγραμμα LIFE είναι 2,5 δις ευρώ για την περίοδο 2007 έως 2013 και εκπροσωπεί μόνο 1,5 του συνόλου των περιβαλλοντικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει σχεδιαστεί ως πλατφόρμα για να αναπτυχθεί η ανταλλαγή καλών πρακτικών και να υπάρξει καταλητική προώθηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, η αποτελεσματικότητα της περιβαλλοντικής συνιστόσα του LIFE είναι καθορίζεται από το κατά πόσον τα χρηματοδούμενα προγράμματα έχουν καταλητικέ επιδράσει στι ε, απαραίτητε αλλαγέ του περιβάλλον. Δεδομένε τη πρόθεση τη Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή να αυξήσει σημαντικά τι δαπάνε για το περιβάλλον στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού, αποφασίστηκε η αποτελεσματικότητα τη περιβαλλοντική συνιστόσα του προγράμματο LIFE να εγκριθεί. Η ακρόαση ε, μάλλον η εξέταση των προγραμμάτων προς χρηματοδότηση οδήγησε στην έγκριση 95 προγραμμάτων που ε, χρηματοδοτήθηκαν από 2007 έως το 2010 σε πέντε κράτη-μέλη μεταξύ των μεγαλύτερων δικαιούχων του Λαιμ Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Συνολικά, το ελεγκτικό συνεδρίο βρήκε ότι το, πρόγραμμα δεν σχεδιάστηκε σωστά και δεν ελοποιήθηκε ακριβώ όπω θα έπρεπε, με αρνητικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητά του. Ποια ήταν τα βασικά προγράμματα, πρώτα απ' όλα, υπήρχαν ε, προβολικά πολλοί στόχοι ε, παρά το περιορισμένο πεδίο του. Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα για το περιβάλλον αφορούν 12 τομεί πολιτική που αφορούν διαφορετικά θέματα και κλάδου, που οδήγησε σε μεγάλη κρίσιμη μάζα καλών προγραμμάτων προκειμένου να υπάρξει αρκετό ανταγωνισμό και σωστή προώθηση τη περιβαλλοντική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που είναι ο πρωταρχικό στόχο του προγράμματο. Επιπλέον, αυτός ο περιορισμένος προπολογισμός περιορίστηκε σε δύο εκμεταμιεύσεις κατά, κατά κρατός μέλος. Εδώ ε, έπρεπε να υπάρξει αναλογική κατανομή των προγραμμάτων μεταξύ των κρατών μελών ε, και αυτό σημαίνει ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων είχαν να κάνουν με την υλοποίηση προγραμμάτων στο ίδιο κράτος μέλος μεν, αλλά όχι με προγράμματα από άλλα κράτη-μέλη. Λόγω των περιβαλλοντικών ωφελών του προγράμματος LIFE θεωρηθεί θεωρήσαμε ότι πρέπει να έχει και μια διάσταση Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο εθνική ώστε ε, τα καλύτερα και ευρύτερα προγράμματα να επιλεγούν εφόσον υπάρξει σωστή υποβολή και ανταγωνιστική διαδικασία για το εθνικό επίπεδο και ωφέλη για το ευρωπαϊκό. Υπήρξαν επικρίσεις για τους δείκτες μέτρησης των αποτελεσμάτων για όλα τα προγράμματα live, οι οποίοι θα έπρεπε κατά καιρούς να συναθρίζονται ώστε να δούμε και τα καλύτερα αποτελέσματα από το κάθε πρόγραμμα. Ο σωστός εντοπισμός των προγραμμάτων ε, επηρέασε την ε, προγραμματισμό την τελική αξιολόγηση η οποία κακώς είναι διαθέσιμη πέντε χρόνια μετά την έναρξη του προγράμματος, δηλαδή δύο ε, χρόνια πριν τη λήξη κάθε προγράμματος. Οι αδυναμίες σχεδιασμού ε, είναι έμφυτες στο όλο πρόγραμμα, οπότε ε, δυσκολεύουν τη σωστή υλοποίησή του ευθύς εξ αρχή. Τα προγράμματα ε, υλοποίηση είχαν τι εξή ελλείψει. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δικαιολογούσε πάντοτε επαρκώ την επιλογή των προγραμμάτων. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερος για την αποτίμηση κάποιων πτυχών που θεωρούνται θεμελιώδεις για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων live ιδίως ο καινοτόμος και αποδεικτικός χαρακτήρας κάποιων ε, στόχων ή οι εκτιμήσεις που έχουν γίνει εκ των προτέρων για τα αποτελέσματα των προγραμμάτων. Το σύστημα επιλογής ενέχει τον κίνδυνο κάποιες πτυχές των προγραμμάτων να μην έχουν αποτιμηθεί σωστά και αυτό να έχει αρνητικέ συνέπειες για τα τελικά τους αποτελέσματα και συνολικά για το κάθε πρόγραμμα δεν δόθηκε επαρκή προσοχή στα πραγματικά αποτελέσματα που επετέχθησαν από το κάθε πρόγραμμα και αυτά τα αποτελέσματα δεν εξετάστηκαν αν μπορούν να είναι μακροχρόνια ή αν μπορούν να ε, εφαρμοστούν κι αλλού. Ένα παράδειγμα, δικαιούχοι ε, οι δικαιούχοι ετοίμαζαν ε, την εκτίμηση και την τελική έκθεση παρουσιάζοντας τις ίδιες τις απόψεις τους για τα επιτεύγματα του κάθε προγράμματος. Το σύστημα παρακολούθησης που εξετάζει το τι γίνεται με τα προγράμματα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, συντάσσει και αυτό από την πλευρά του κάποιες εκθέσεις. Οι δικαιούχοι έχουν κάποια φυσική τάση να είναι υπερφιλόδοξοι όταν εξετάζουν τα επιτεύγματα του κάθε προγράμματός τους και γίνονται πολλές δηλώσεις από τους ίδιου, που απλώς ε, Της αντιγράφει η ομάδα παρακολούθησης την έκθεση που συντάσσει. 72% των προγραμμάτων τελικά δεν πέτυχαν τα αρχικά τους αποτελέσματα και ε, το ίδιο και από, τις, από τους ελεγκτές ε, του συστήματος παρακολούθησης που ε, υπερτίμησαν τις δυνατότητες του κάθε προγράμματος. Όπως είπα προηγουμένως, ένα από τα προγράμματα, ένα από τους βασικούς στόχους του προγράμματος LIFE είναι να έχει καταλητική επίδραση στην ανάπτυξη της ε, περιβαλλοντικής πολιτικής και των περιβαλλοντικών δράσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι τα αποτελέσματα των προγραμμάτων να διαδίδονται επαρκώς και σωστά και να ε, αξιοποιούνται. Αυτό δείχνει παρόλα αυτά ότι έχουμε ακόμη κενά σε αυτή τη διαδικασία. Ακόμη και όταν τα στηριζόμενα προγράμματα έχουν πετύχει θετικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα, τα προγράμματα δεν καταλήγουν να διαδίδονται σωστά, ούτε να αξιοποιούνται και έτσι αυτά τα μικρής κλίμακας αποτελέσματα δεν έχουν αξία για την κλίμακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, οι δικαιούχοι προγραμμάτων που είναι ιδιωτικέ εταιρείε πολλέ φορέ έχουν προγράμματα με στατηγικό ε, πλεονέκτημα. Και προκειμένου να προστατευτεί η τεχνογνωσία του, οι διαδικασίε ε, διάδοση συνδέονται με εμπορικέ δράσει που δεν συμπεριλαμβάνουν συνολική περιγραφή του προγράμματο. Αυτό ε, μειώνει σοβαρά την δυνατότητα αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματο και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Έτσι, μόνο 8 από 23 ολοκληρωμένα προγράμματα που έχουμε εξετάσει ε, είτε αξιοποιήθηκαν είτε πρόκειται να αξιοποιηθούν. Αυτό κατά την άποψή μου δεν είναι καλό αποτέλεσμα. Το συνέδριο επίση στην έκθεσή του συμπεριλαμβάνει κάποιε συστάσει, οι οποίε σκοπό έχουν να καλύψουν όλα αυτά τα θέματα και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τη περιβαλλοντική συνιστόσα του προγράμματος LIFE. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να περιορίσει την ε, επιλεξιμότητα των ε, δικαιωχών και να ορίσει ε, μια διάρκεια ετών, ώστε να επιγραμμιστεί η διαδικασία επιλογή και να επικεντρωθεί ε, σε συγκεκριμένα ζητήματα καθώς και την αξιολόγηση τη της διάστασης του προγραμματισμού. Επίσης πρέπει να βεβαιωθεί ότι τα προγράμματα επιλέγονται βάσει της αξίας τους και της γεωγραφικής τους ε, εμβέλειας και επίσης να μην διαταράσσεται η ίση η ε, προσφορά ίσων ευκαιριών μεταξύ των χωρών. Επίσης θα πρέπει οι αξιολογητές να προβλέπουν ξεχωριστή βαθμολόγηση και καταχώρηση των αποτελεσμάτων ανάλογα με, τα, ε, με τους αρχικούς στόχους των δικαιούχων και τις προτάσεις τους, καθώς και να υπολογίζουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων στο μέλλον. Θα πρέπει να εισαχθούν δείκτες ε, για τα αποτελέσματα, κοινοί δείκτες για τα αποτελέσματα, προκειμένου να γίνεται σωστά η διαδικασία παρακολούθησης των προγραμμάτων. Επίσης η ομάδα παρακολούθησης θα πρέπει να οργανώσει σωστά την αποτίμηση, αλλά, τόσο, αλλά και τη διάδοση των αποτελεσμάτων και για άλλους δικαιούχους. Και στη δική της έκθεση παρακολούθησης κατά την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος με τις ε, επισκέψεις εκπόστη. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε επίσης την διάδοση και την, ε, βελτίωση των, την καλύτερη μετάδοση των αποτελεσμάτων των ιδιωτών δικαιούχων, ακόμη και με εμπορικέ δράσει. Αυτή ήταν η εισηγησή μου. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και είμαι για διάθεσή σα. Σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κίνηση, και δίνω το λόγο στην εισηγητρία Γιούτα Χάουκ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Η έκτακτη έκθεση της, ε, του ελεγκτικού συνεδρίου είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Η συγκεκριμένη αυτή όμως έκτακτη έκθεση αφορά την υλοποίηση του LIFE και την αξιολόγηση από το ελεγκτικό συνέδριο των αποτελεσμάτων αυτής της υλοποίησης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με νομοθεσία γνωστή και καλούμεθα να την αξιολογήσουμε αλλά με μεγάλη καθυστέρηση. Θα έπρεπε αυτό να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Εμείς ήμασταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για το αποτέλεσμα των ε, προσπαθειών μας σε συνεργασία με την Ιρλανδική Προεδρία. Και θα θέλαμε να είχαμε προχωρήσει πολύ νωρίτερα ώστε να μην φτάσουμε μέχρι τώρα τον Απρίλιο να γίνει η πρώτη προκήρυξη. Εφόσον ήμασταν από τα μέσα του έτους ε, πέρσι έτοιμοι να κλείσουμε το νομοθετικό έργο. Κατά τα άλλα πάντως είμαι υπερήφανη, πρόεδρε, διότι έχουμε τουλάχιστον κερδίσει σε ένα πεδίο τον αγώνα για τα ολοκληρωμένα προγράμματα, γιατί ήμουν εξ αρχής υπέρ αυτής της προσέγγισης. Και ναι, μπορεί να έχουμε κάποια άλλα παραδείγματα ολοκληρωμένων προγραμμάτων, τουλάχιστον όνομα ολοκληρωμένων προγραμμάτων, το Λούξ επί παραδείγματι για την Ιβυρική, το ελεγκτικό συνέδριο όμως θα έπρεπε ίσως μέσα σε δύο χρόνια να έχει έτοιμη την προσεχή έκτακτη του για να μας θέσει και αυτά να τα αξιολογήσουμε. Αυτά τα οποία επικρίνει ο κύριος Κίνστ έχουν να κάνουν με τις εθνικές πιστώσεις και τις επικρίσεις ως προς την αξιοποίησή τους. Είναι κάτι το οποίο και εμείς το βλέπουμε το έχουμε υπογραμμίσει, μια ομάδα τουλάχιστον από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι θα έπρεπε να διατυπώνεται ή να διαμορφώνεται η χρήση αυτών των εθνικών πιστώσεων κατά τρόπον ώστε να προβάλλεται πολύ περισσότερο το έργο και η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πρόκειται για ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό θα πρέπει να το δούμε με μια σταδιακή μείωση των εθνικών πιστώσεων. αλλά τα κράτη-μέλη θέλαν να διατηρήσουν επαόριστον μάλιστα τις εθνικές πιστώσεις. Εν πάση περιπτώσει καταφέραμε εμείς να περάσουμε την πρόταση για τη σταδιακή μείωση και εξαφάνισή τους. Για την ε, δυνατότητα επανάληψης θα ήθελα να είχαμε κάποιους φορείς όπου να, οι, για, οποίοι είναι σε θέση, προγράμματα τα οποία έχουν λειτουργήσει καλά σε ένα κράτος μέλος και θα μπορούσαν αντίστοιχα έστω και με άλλες συνθήκες και προϋποθέσεις να ε, μεταφερθούν σε ένα άλλο κράτος ή εν πάση περιπτώσει να αξιοποιήσουν τα διδάγματα της πρώτης υλοποίησης στο άλλο κράτος μέλος, να το συντονίζουν αυτό. Θέλαμε δηλαδή ένα είδος δικτύου μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών των αρχών δηλαδή οι οποίες εργάζονται για το LIFE. Πράγμα το οποίο θα είχε ε, τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει και το ρόλο της, ε, τον παιδευτικό των υπηρεσιών εκείνων οι οποίες ε, όταν πια δεν θα υπάρχουν οι εθνικές ε, πιστώσεις θα είναι σε θέση, θα έχουν μάθει πώς να διαχειρίζονται τα κονδύλια αυτά. Το πρόγραμμα εργασίας, όπως θα το αποφασίσει και η Επιτροπή με το Συμβούλιο και η δική μας ε, Επιτροπή, θα πρέπει να το αντικατοπτρίζει αυτό. Και έχω και ερώτηση προς την Επιτροπή εν προκειμένου σε ποιο βαθμό για το τρέχον πρόγραμμα live από το 14 έως το 20. Σε ποιο βαθμό λοιπόν έχει λάβει υπόψη, έστω και όταν ε, είχε πια κλείσει η νομοθετική διαδικασία, ε, παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου για να προσαρμόσει αντίστοιχα το πρόγραμμα εργασίας της. Και αυτό όχι μόνο για τις προτεραιότητες, αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας των μέσων και τις διαδικασίες επιλογής. Εσείς, παραδείγματι, επικρίνατε το σύστημα της, ε, ή το μηχανισμό αξιολόγησης στις επιλογές. Υπάρχει κάτι καινούριο Υπάρχει μια ε, διαφορετική λύση για το πώς μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα ή πώς μπορεί ένα έργο το οποίο έχει υλοποιηθεί να αξιοποιηθεί ως υπόδειγμα ή ως παράδειγμα για κάποια άλλα έργα. Και πώς μπορείτε κι εσείς ε, να βοηθήσετε στο να αναπτυχθεί ο καταλυτικός ρόλος, ρόλος καταλήτη ενός έργου, το οποίο έχει σωστά και καλά αξιοποιήσει τα ε, ευρωπαϊκά κονδύλια, τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Φορολογημένου τελική αναλύση, ώστε να αναπτυχθούν έργα για την προστασία του περιβάλλοντος. Και θα ήθελα για τον κύριο Κίνς να κάνω την εξή ερώτηση. Το τωρινό ε, πρόγραμμα LIFE, ο τωρινό του προπολογισμό, λέτε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί. Άλλωστε το έχει προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτό. Προβλέπετε μια αύξηση, όχι στο βαθμό που θα θέλαμε όλοι. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια αύξηση και φαίνεται ότι αυτή η αύξηση αφορά μόνο το νέο κομμάτι, δηλαδή την ε, πολιτική για τις κλιματικές αλλαγές, για το κλίμα. Έχω λοιπόν την έξω ερώτηση. Με τη δική σας ανάλυση κύριε Κίνστ, γιατί αναφερθήκατε στην ε, πολιτική για το περιβάλλον και την πρακτική της υλοποίησης από τη διοίκηση. Στο βαθμό λοιπόν που εξετάσατε όλες αυτές τις διαστάσεις, τι είδους διδάγματα μπορείτε να αντλήσετε για το κομμάτι που αφορά την πολιτική για το κλίμα στο νέο πρόγραμμα. Και πάνω απ' όλα, εκεί όπου αναφέρεστε στο γεγονός ότι δεν ήταν αρκετά καλά εστιασμένα τα έργα με, το, με τα νέα ε, δημοσιονομικά μέτρα που πρόκειται να προταθούν στο, ή μέσα καλύτερα, τα νέα δημοσιονομικά μέσα που πρόκειται να προταθούν στο τμήμα που αφορά την κλιματική πολιτική, ε, σε αυτή την ε, φάση και από αυτή του τη θέση το ελεκτικό συνέδριο τι άλλο θα μπορούσε να προτείνει συγκεκριμένα. Έχετε κάποιε υποδείξει ενδεχομένω για την Επιτροπή και για την υπηρεσία, την αποκεντρωμένη υπηρεσία που αναλαμβάνει την εκτέλεση. Ώστε να τις δούμε από τώρα και να μην περιμένουμε σε δύο-τρία χρόνια να δούμε εκ των υστέρων ε, ε, κριτική. Θέλουμε τώρα, την ώρα που αρχίζει η υλοποίηση, να ε, ξέρουμε πού εντοπίζονται τα προβλήματα και οι προτάσεις. Θα ήθελα επίσης για την ομάδα ε, παρακολούθησης, monitoring team, που έχετε, να ρωτήσω το εξής. Αναφερθήκατε στην monitoring team τόσες φορές. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Επιτροπή? Εκπρόσωποι κρατών μελών? Υπάλληλοι? Ποιοι είναι αυτοί που απαρτίζουν την ομάδα παρακολούθησης? Και ρωτώ γιατί δεν είμαι μέλος μόνο εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και εισηγήτρια για το πρόγραμμα LIFE. Είμαι και στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών και ασχολούμαι πολύ με τους προϋπολογισμούς και βλέπω ότι έρχεται ένας όγκος και απαιτήσει εργασίας ε, σημαντικός ή ίσως όχι, δεν ξέρω, δεν θέλω να, προδικάσω τίποτα ή μπορεί να είναι και περιορισμένο αυτή η επιβάρηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης από κάπου πρέπει να πληρωθούν. Ερωτώ λοιπόν εσείς, τι θεωρείτε, θα πρέπει να, προσ... να καλύψει τους μισθού τους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, ε, πώ θα λειτουργήσει αυτή η ομάδα εργασία, η ομάδα παρακολούθησης. Δεν έχουμε και πολλούς συναδέλφους που διατυπώνουν ερωτήσεις εδώ από την Επιτροπή μας, αλλά νομίζω ότι οι πιο αξιόλογοι είναι παρόντες. Ούκεν το πολλό το F, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Γεμπράντη. Yes, Utah, thank you. είχαμε πει θα πρέπει να πούμε ότι επικρίνεται εσείς το Συμβούλιο, όπως άλλωστε και εμείς, ή ότι χρειάζονται περισσότερα χρήματα κτλ. Το Συμβούλιο όμως, τα κράτη-μέλη, θέλουν στο δυνατόν περισσότερους στόχους. Γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούν να βρίσκουν λύσεις για να αξιοποιούν κονδύλια στις χώρες τους. Επίση επικρίνεται τις εθνικές πιστώσει. Μα αυτό ήταν μια από τι μεγαλύτερες μάχες που είχαμε με το Συμβούλιο. Και είναι γελίο να έχουμε με το live τέτοια προβλήματα. Θα έπρεπε να έχουμε πετύχει σταδιακή μείωση των εθνικών ε, μεροδοτήσεων. Ή να μην υπάρχουν και καθόλου. Αυτή αυτό είναι το βασικό μου μήνυμα. Πώς το μήνυμα όμως αυτό θα περάσει στα κάτι μέλη, αυτό είναι το ερώτημα. Εκεί είναι το σοβαρότερο πρόβλημα. Στην έκθεσή σα απευθύνεστε επανελειμμένο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ νομίζω θα πρέπει να κεντρωθούμε ακόμη περισσότερο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα τα κράτη-μέλη. Και τελευταία μου παρατήρηση και εδώ να στηρίξω και να συμφωνήσω με την Γιώτα Χάουκ. Εδώ μιλάμε για την περίοδο 2005-2010. Νομίζω το 2011 όμως ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με το πρόγραμμα LIFE εδώ στο σώμα μας. Θα ήταν ε, πραγματικά πολύτιμο, ε, εξαιρετική σημασία μάλλον έχουμε, την έκθεση αυτή πριν αρχίσουμε να εργαζόμαστε. Διότι όλα τα επιχειρήματα που χρησιμοποιείται Είναι επιχειρήματα που και εμεί χρειάστηκε να προβάλλουμε στου τριμερεί διαλόγου με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Και δεν είναι μόνο αυτή η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που αφορά το πρόγραμμα, αλλά έχω δει κι άλλε το τελευταίο δίμηνο που αφορούν την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Θα ήταν λοιπόν πολύ χρήσιμο για μα ω Κοινοβούλιο στις ε, σε ζητήσει μα και στι εξοπλισμούς μα με το Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τώρα την, ε, το χρονοδιάγραμμα, νομίζω το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για το ερχόμενο διάστημα καλύπτει μια επταετία. Έχουμε και μια ενδιάμεση όμως έκθεση το 2016. Μπορεί να βρεθούν τρόποι να ξεκινήσει αξιολόγηση της ε, τρέχουσας περίοδου προγραμματισμού εγκαίρως ώστε τα πρώτα σας πορίσματα να τα χρησιμοποιήσουμε για το 2016 και την ενδιάμεση έκθεση. Ίσως με κάποιες σύντομες διαδικασίες να γίνεται αυτό για την ενδιάμεση έκθεση του 2016. Όχι μόνο για το live, αλλά και για άλλα εργαλεία που μας αφορούν. Νομίζω θα ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικό. Όπω θα έπρεπε να προβλέψει το Ελληνικό Συνέδριο για την τωρινή περίοδο του πολιτέ δημοσίου πλαισίου. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλημέρα σα. Ήδη ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε θετικά στην έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου. Ορισμένα θέματα τα έθεσε και η συγγήτρια Γιούτα Χάουκ. Οι βασικέ ιδέε τη έκθεση, δηλαδή ουσιαστικά αντικατοπτρίζονται και στο νέο κανονισμό για το πρόγραμμα LIFE, που ξέρετε ότι αποτέλεσε αντικείμενο έντονων συζητήσεων μεταξύ Κομισιών και Συμβουλίου. Θα ήθελα εδώ να τονίσω το γεγονό ότι σε ό,τι αφορά τι εθνικέ εισφορέ, ε, για τι οποίε ασκείται έντονη κριτική, ε, στην ενδιάμεση αξιολόγηση σταδιακά θα μειωθούν μέχρι να εξαλειφθούν. Και υπήρξαν και άλλα θέματα που αφορούσαν τη νομική βάση. Έχουμε τώρα μεγαλύτερη εστίαση του προγράμματος Live θα τα δείτε και στην ενδιάμεση αξιολόγηση. Θα ήθελα να μιλήσω για κάποιους νεοτερισμούς τώρα, διότι το νέο πρόγραμμα LIFE δεν αποτελεί αντιγραφή, επικόλυση ε, του προηγούμενου. Γιατί είπε και ο κύριος Κίνστο ότι πρέπει να έχει ρόλο καταλήτη αυτό ε, το πρόγραμμα LIFE και με βάση και την πρικοδότησή του ίσως να μην μπορεί να τα καλύψει όλα. Αυτή η έννοια λοιπόν των ολοκληρωμένων προγραμμάτων ε, είναι μια θετική έννοια για να μπορέσει να συνεχίσει να διδραματίζει ρόλο καταλήτη το πρόγραμμα LIFE αλλά και για να βελτιωθεί το επίπεδο εφαρμογής και του περιβαλλοντικού πλαισίου. Γνωρίζετε ότι πρέπει σε διάφορους τομείς ε, να σημειωθεί πρόοδος όπως είναι η ποιότητα των υδάτων, του αέρα, και θέλουμε να εξασφαλίσουμε τα κονδύλια να χρησιμοποιούν τουλάχιστον κατά τρόπο ώστε ορισμένε χώρε που αντιμετωπίζουν δυσκολίε στην εφαρμογή να ε, βοηθηθούν για να αξιοποιήσουν ω ε, το δυνατόν περισσότερο το πρόγραμμα και να αξιοποιήσουν τα κονδύλια και άλλων ε, ταμείων. Γιατί ξέρετε ότι και σε άλλου τομεί, όπω παραδείγματο χάρη στην πολιτική συνοχή, διατίθεται κονδύλια και από αλλού. Πρέπει να αξιοποιηθούν όλα αυτά. Επαναλαμβάνω ότι εμείς θα επικεντρωθούμε και στο κλίμα και στα απόβλητα και στην ποιότητα του αέρα και των υδάτων. Μια άλλη καινοτομία. Ξέρετε ότι συζητάμε στα κράτη-μέλη, στο πλαίσιο του πρώτου πολιετούς προγράμματος εργασίας, υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που δυσκολεύονται να δεχθούν ε, κάποιες έννοιες για αυτό το πρόγραμμα LIFE, αλλά η πιλωτική φάση έχει εγκριθεί, έχει ξεκινήσει και έτσι θα μπορέσουμε να δούμε αν μπορεί να λειτουργήσει, ιδίω ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματος και για τη βιοπικιλότητα. Και με τη νέα νομική βάση νομίζω ότι θα μπορέσει το ΛΑΒ να έχει καταλητικό ρόλο και να βελτιωθεί και η εταιρική σχέση δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Άρα να είναι πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό το πρόγραμμα. Να τονίσω επίσης ότι έχουμε ένα νέο σκέλος ε, ενημέρωσης και επικοινωνίας. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα μπορούν κατά κάποιο τρόπο να εφαρμόζουν ε, με τον ίδιο τρόπο το ε, ρυθμιστικό πλαίσιο και θα μπορούν να εφαρμόζονται πρωτοβουλίες για τη διαδικτύωση και για την ανταλλαγή εμπειριών χώρες δηλαδή που έχουν θετικές εμπειρίες να βοηθούν λιγότερο προηγμένες στην εφαρμογή του LIFE χώρες. Το LIFE θα είναι πιο κοντά στις πολιτικές και θα λαμβάνει υπόψη το περισσότερο, ε, μάλλον θα λαμβάνονται περισσότερο και σε άλλες πολιτικές περιβαλλοντικές ε, πτυχές. Πρόεδρος, να δώσω στην Σαντρίν Μπελίε και όποιον άλλο συνάδελφο στη συνέχεια επιθυμεί το λόγο. Κυρία Μπελίε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κίνστ για την παρουσία του αφενός και για την έκθεση των αποτελεσμάτων του, του Ενεκτικού Συνδρού το πρόγραμμα LIFE λοιπόν που όπως υπενθύμισαν οι συνάδελφοι είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς όμως είναι μια μικρή σταγόνα στον ωκεανό, στο πλαίσιο δηλαδή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Μια σταγόνα που, αν δει κανεί ε, τη δουλειά που έχει κάνει το κοινοβουλίο μας και ιδίω ε, συγκεκριά μας για το θέμα αυτό, είχαμε μια αύξηση, θα τη θέλαμε μεγαλύτερη βέβαια, είχαμε πάντως μια αύξηση του προϋπολογισμού, καλοδεχούμενη, και είχαμε και έναν επαναπροσανατολισμό δηλαδή να καταπολεμηθεί η απώλεια της βιοπικιλότητας που όλο και πιο αισθητή γίνεται ε, ο στόχος. Σε ό,τι αφορά το ίδιο το πρόγραμμα, το είπαν και οι συνάδελφοι, με τα συμπεράσματά μας ε, ενισχύονται οι πεπιθήσεις, η πεποίθηση τουλάχιστον η δική μου ότι χρειάζεται βερετέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας, υπάρχουν περιθώρια, έχετε προτείνει διάφορα μέτρα, λυπούμε όμως που δεν είχαμε τα συμπεράσματα αυτά νωρίτερα, πριν δηλαδή τις συζητήσεις σε σχέση με το νέο πρόγραμμα LIFE. Δεν αποκλείω βέβαια το να υπάρξει δυνατότητα στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία να εξετάσουμε το ενδεχόμενο αναθεώρησης. Μεταξύ των προτάσεων για βελτίωση σημειώνω καλύτερη στόχευση των χρηματοδοτικών έργων και προγραμμάτων και να είναι μετρήσιμα, όπως λέτε, να είναι παρκώς ορατά, να έχουν την προβολή που απαιτείται ώστε να μπορούν να υπάρχει αυτή η επανάληψη, αυτή η αντιγραφή. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τις απαιτήσει, υπάρχουν και οικολογικές ε, παράμετροι με τις οποίες συμφωνούμε. Δύο ε, θέματα έχω να θέσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτο, βούληση της Κομισιόν να εγκρίνει το πρόγραμμα περί αποζημίωσης για περιβαλλοντικά θέματα. Μια χήμερα είναι μέχρι στιγμής αυτό. Ε, γιατί ξέρουμε ότι αν ένα οικοσύστημα καταστραφεί δεν μπορεί να ανασυσταθεί, αλλά μας απασχολεί πάρα πολύ και η ανάγκη, οι απαιτήσει που υπάρχουν και μας το λένε και οι τοπικοί παράγοντες για τοπική χρηματοδότηση, για τη διατήρηση ε, των φυσικών χώρων και χρηματοδότηση του LIFE για τη διατήρηση των φυσικών χώρων. Νομίζουμε ότι ανταποκρίνεται στη γνωστή κατ' εμά ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή υλοποίηση οδηγίας για τα ενδιατήματα και για τα πτηνά. Μέτρα αποζημίωσης λοιπόν, αντιστάθμισης, είναι ένα θέμα, είναι ένα ερωτηματικό. Και το ερώτημά μου κυρίως είναι η επιλογή ε, απόδοσης των κονδυλίων με ποιες ε, παραμέτρους αποφασίζεται και ποια είναι η πολιτική αντιστάθμιση αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας βιοπικιλότητας. Σε ό,τι αφορά τώρα τη χρηματοδότηση αυτή και την απώλεια της βιοπικιλότητας, σε ποια κοινωτική πολιτική στηρίζεται και αν ελεκτικό συνέδριο και κομισιόν θεωρούν ότι αποτελεί καλή χρήση του προπολογισμού αυτού που ήδη είναι περιορισμένος. Δεύτερο ερώτημα το είδος ε, της χρηματοδότησης που προβλέπει η Κομισιόν ε, για τον περιπολισμό LIFE, για το κλίμα συγκεκριμένα, για αυτό το πρόγραμμα. Η επιτυχία του LIFE, όπως υπενθυμίσατε κι εσείς, βασίζεται στο κατά πόσον μπορεί να χρηματοδοτεί πιο πολύ ε, μέτριας κλίμακας προγράμματα, που όμως έχουν αισθητή, ορατή επίδραση στο περιβάλλον. Όμως η γάμα δέλτα κλίμα λέγεται ότι θέλει να χρησιμοποιήσει 80 εκατομμύρια ευρώ για την ε, συγκέντρωση πόρων σε ιδιωτικέ τράπεζες. Ισχύει αυτό και πώς αιτιολογεί τη χρήση του προπολογισμού και αυτού του κομματιού του προπολογισμού του ΛΑΕΦ για αυτό το στόχο. Εσείς τι άποψη έχετε για μια τέτοια χρήση του προπολογισμού ΛΑΕΦ, κύριε Κίνστ. Η κυρία Λούμπιτσεβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένη με αυτή την έκθεση και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κίνστ και την ε, Γιούτα για όσα είπαν. Ως προς την αξιοποίηση του προγράμματος LIFE. Το, το πρόγραμμα αυτό το βρίσκω πολύ χρήσιμο, αν και δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στη δική μου τουλάχιστον τη χώρα. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτή την έκθεση και σε επίπεδο κρατών μελών. Είναι σημαντικό να λάβουμε εθνικά μέτρα για τη βελτίωση της συμμετοχής των κρατών μελών στο πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προβλέψουμε μέτρα για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η, ε, η, τα, η αποδοτικότητα του προγράμματος. Ακούσαμε σήμερα ότι υπάρχουν ελλείψεις ως προς αυτή τη διάσταση. Σε κάποια κάτι μέλη υπάρχει πεποίθηση ότι το πρόγραμμα LIFE και τα κονδύλια του είναι κάτι το μοιραίο το αναπόφευκτο. Είναι κάτι δηλαδή που το θεωρούν λίγο δεδομένο ε, και έτσι δεν γίνεται τίποτα για την ποιότητα του προγράμματος. Υπάρχει κάποια στατιστική ανάλυση, μελέτη για τα κράτη-μέλη για τα οποία το πρόγραμμα αυτό είναι πιο χρήσιμο ή μάλλον που απορροφούν καλύτερα και αξιοποιούν τα κονδύλια. Δεν μιλάω για να κατονομάσουμε ή να απενοδίσουμε τους ε, κακούς μαθητές, αλλά να βρούμε τρόπους να ενθαρρύνουμε τους μέτριους μαθητές να βελτιώσουν τους βαθμούς τους. Γι' αυτό νομίζω ότι κάποιες σχετικές πληροφορίες θα ήταν χρήσιμες για να τις αξιοποιήσουμε και στα κρατημέλη. Και εν τέλει Ευχαριστώ για τα σχόλια και τις αντιδράσεις. Θα ήθελα ξεκινώντας να πω ότι και εγώ είμαι από τους ε, υποστηρικτές του προγράμματος FAN, από τους FAN του προγράμματος LIFE και Γι' αυτό χάρηκα πολύ ε, για τη δυνατότητα που υπάρχει. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με τα σχόλια της κυρίας Χάουκ. Καταρχάς, η, χρονική, ο χρονισμός αυτής της έκθεσης, η χρονική σύμπτωση. Βεβαίω, αν μπορούσαμε να διπλασιάσουμε τον αριθμό των απασχολημένων πριν το τέλος μιας προγραμματικής ε, περίοδου και να έχουμε διακοπές στην πρώτη διετία μετά την ε, ολοκλήρωση ενός προγράμματος ε, και πριν την έναρξη τη επόμενη προγραμματικής περίοδου, θα καταφέρναμε να κάνουμε και πιο νωρί εκθέσεις μα. Αλλά ξέρετε έτσι είναι η δουλειά που μα πέφτει με τα προγράμματα όπω εξελίσσονται. Κάνουμε ό,τι μπορούμε στο μέγιστο των δυνάμεών μα εργαζόμαστε και ο κύριο Γερμπράντη που ξέρει καλά το ελεκτικό συνέδριο ασφαλώς αντιλαμβάνεται ότι καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Ελπίζουμε να βελτιωθούμε βέβαια. Πάντω. και με τη δημοσίευση αυτής της εκθέσεως στα μέσα Ιανουαρίου του 2014 έστω και με αυτή την ε, καθυστερημένη δημοσίευση κάνουμε ό,τι μπορούμε διότι δεν μπορούν όλα να μεταφραστούν, να μεταφερθούν στο κύριο νομοθέτημα πολλές από τις ε, παρατηρήσεις μας έχουν να κάνουν με τη δευτερογενή νομοθεσία, καλύτερα τις πράξεις εκτελεστικές, κατεξουσιοδότηση λοιπά. Συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν να κάνουν με τα λειτουργικά μέσα που μπορούν ε, να αξιοποιηθούν. Και τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα τα είχαμε διαθέσει στην Επιτροπή ε, στα μέσα του 2013 και έτσι πιστεύω ότι ήταν γνωστές οι τάσεις ή τι άλλο της εκθέσεως. Εν τέλει, και πριν από πέντε χρόνια είχαμε δημοσιεύσει την ειδική έκθεση για μια άλλη πτυχή του προγράμματος Life, το Life Nature, που δεν είναι βέβαια το ίδιο με το Life Environment, με το Life για το περιβάλλον, αλλά πάντως υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με τη διάδοση, με την επικάλυψη, με την εφαρμογή, που σχετίζονται και μπορούν να βρουν αντίκτυπο, ε, απίκηση καλύτερα και σε αυτήν εδώ την έκθεση. Είναι ενθαρρυντικές οι ενδείξεις που έχουμε από τις αρχές της εκτέλεσης. Πάντα είμαστε επιφυλακτικοί βεβαίως, αλλά πάντως βλέπουμε ένα καλό εργαλείο συνεργατικής ε, ε, δράσης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των ε, εθνικών πιστώσεων ή κοινοτικών. Το ολοκληρωμένο λοιπόν πρόγραμμα είναι ένα καλό μέσον και ελπίζουμε ότι θα δούμε να λειτουργούν όλο και πιο αποτελεσματικά με την ολοκλήρωση αυτή σε περιφερειακό, εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αυτό βασικά σημαίνει το live. Για τις εθνικές πιστώσεις. Από ό,τι βλέπω όλοι συμφωνούμε, ούτε το Κοινοβούλιο, ούτε η Επιτροπή, ούτε το ε, συνέδριο, το ελεγκτικό συνέδριο ήταν υπέρ των εθνικών πιστώσεων. Πλην όμω για το πρώτο ήμιση αυτού του κανονισμού, στην πρώτη προγραμμα... στο πρώτο κομμάτι δηλαδή, τη προγραμματική ε, περίοδου, θα έχουμε αυτό το σύστημα των εθνικών πιστώσεων. Είναι δυνατόν να το διαχειριστούμε σωστά, εφόσον ληφθούν υπόψη και όλε οι άλλε πτυχέ των συναφών άρθρων του κανονισμού. Όπου, εάν τα διαβάζω σωστά, δεν είναι ορθό ένα κράτο μέλο τα χρήματα αυτά να τα εισπράττει, εφόσον δεν είναι σε θέση να παράσχει επαρκό, επαρκούς ποιότητας προγράμματα. Είναι με παρακολούθηση διαχείριση αυτών των δαπανών, αλλά πρέπει να είναι αυστηρή η στάση της Επιτροπής. Και εφόσον ένα κράτος μέλος δεν είναι σε θέση να υποβάλει έργο, το οποίο να είναι ανταγωνιστικό σε αντίστοιχα, στη σχέση με αντίστοιχα έργα που έχουν υποβάλει τα άλλα κράτη-μέλη, τότε έχουμε μόνο την εθνική, την ενδεικτική εθνική πίστοση και όχι την ε, σταθερή ή συγκεκριμένη εθνική πίστοση που εφαρμόζεται. Αυτό είναι ένα τρόπο να ελεγχθούν να είναι των προβαλλωμένων έργων. Και ξέρετε ότι αυτό και ο κανονισμό προβλέπει ότι υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, το capacity building μεταξύ των κρατών μελών που ενδεχομένω έχουν χαμηλή δυνατότητα απορρόφηση. Είναι μια πολύ καλή υποστήριξη, ένα μηχανισμό υποστήριξη όπου δεν μπορεί κανεί να ισχυριστεί ότι έχει αφαιθεί στη μοίρα του και δεν έχει καμία βοήθεια από του άλλου. Όχι. Είναι, εν πάση περιπτώσει, ένα συμβασμό μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου μπορεί και να, να λειτουργήσει καλά. Έχουμε αρκετή εμπειρία, πιστεύω, και σε επίπεδο κρατών μελών για το, από το πρώτο πολίτες ε, πρόγραμμα εργασίας ώστε να αξιοποιηθεί και για το δεύτερο κομμάτι ε, του κανονισμού όπου θα έχουν ε, τελείως εξαλειφθεί οι εθνικές πιστώσεις. Η επικάλυψη, η επανάληψη ήταν ένα ζήτημα για μας, το αναφέρατε και πολλοί από εσά ότι αποτελεί ένα σημαντικό σημείο που μπορεί να χρειάζεται προσοχή στον κανονισμό αυτό. Είναι κάτι το οποίο και εμείς έχουμε εντοπίσει. Πρέπει δηλαδή να αξιοποιηθεί ως καταλήτης για αλλαγές, περιβαλλοντικές αλλαγές, αλλαγές στις πολιτικές για το περιβάλλον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από τη δική μου τουλάχιστον αντίληψη και την παρατήρηση της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου, εδώ έχουμε περισσότερο να κάνουμε μια προσέγγιση από τη βάση και προς τα άνω και όχι άνωθεν. Δηλαδή ορίζονται οι κύριε προτεραιότητε έχουμε ανάγκη από ένα επαρκή όγκο, μάζα έργων που μπορούν να επαναληφθούν και δεν έχουν αποκλειστικά εθνικό ή ακόμα περισσότερο ε, τοπικό χαρακτήρα και μπορούν να επαναληφθούν κάπου αλλού. Εγώ για τις ελεκτικές αυτές αρμοδιότητες που έχουμε επισκέφθηκα δύο, σε δύο περιπτώσεις έργα και ήταν καθαρό για μένα το πώς μπορούν να έχουν καταλητική δράση για ευρύτερες αλλαγές και ακόμα για την περιβαλλοντική πολιτική μιας χώρας. Έστω και ένα μεμονωμένο πρόγραμμα ε, όπου πληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις για τη διάδοση κτλ. Και δεν είχα την εντύπωση ότι στο σχεδιασμό του προγράμματος θα μπορούσε να υπάρχει ενδιαφέρον για τη διάδοση. Και δεν ε, επέτυχαν έτσι. Από τα 23 προγράμματα, τα 8 μπορεί να επαναληφθούν από ό,τι βλέπουμε. Δεν είναι τόσο καταπληκτικό αυτό το αποτέλεσμα για μένα, παρότι η Επιτροπή λέει ότι σε καινοτόμα προγράμματα δεν μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό επανάληψή. Φυσικά δεν είμαστε αφελεί και να περιμένουμε ότι το 100% αυτών των καινοτόμων προγραμμάτων θα επαναληφθεί, αλλά των έργων θα επαναληφθεί, αλλά ένα στα τρία είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Προπολογισμό. Στην έκθεση και ήταν μάλιστα μια από τις πρώτες μας συστάσεις. Είχαμε όντως επισημάνει αυτή την έλλειψη ισορροπίας μεταξύ πολύ περιορισμένου ή σχετικά περιορισμένου προϋπολογισμού, πρικοδότησης και πολύ υψηλών φιλοδοξιών. Εμείς ο λεκτικό συνέδριο είμαστε προσεκτικοί και δεν διατυπώνουμε κρίσεις για το ε, δημοσιονομικό πακέτο, δεν ε, θέλουμε να υψέλθουμε στην επιλογή την πολιτική που ανήκει στο νομοθέτη για το πόσο θα χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμα, αλλά με ενίσχυση αυτής της φιλοδοξίας σε σχέση με το παλαιό πρόγραμμα LIFE δεν μπορούσε να λειτουργήσει καλά το πρόγραμμα με περιορισμένο προϋπολογισμό Με μία μόνο προκήρυξη για υποβολή προτάσεων σε μία χώρα και μία προτεραιότητα μόνο ή ένα τομέα προτεραιότητας ε, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί επαρκή χρηματοδότηση. Άρα βλέπαμε ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα του ανταγωνισμού. Σε αυτό επικρίνουμε, ότι δεν έχει περιθώριο για ανάπτυξη ανταγωνισμού μεταξύ των προτάσεων και των έργων. Αλλά είναι προφανές, δεν μπορούμε να έχουμε... Ε, δεν μπορούμε να παίζουμε σε πολλές ορχήστρες όταν δεν έχουμε αρκετά λεφτά, όπως λέμε στα τσέχικα. για τις πιστώσεις ε, και το κλίμα θα αφήσω τα σχόλια στους συναδέλφους. Για την ομάδα επιτήρησης δεν θα σχολιάσω εγώ, δεν είμαι αρμόδιος για να πω ποιος θα συμμετάσχει. Από την άλλη βέβαια επικρίνουμε συγκεκριμένα ζητήματα που δεν παρακολουθούν οι ομάδες, δηλαδή ζητήματα που έχουν να κάνουν και πρέπει να ληφθούν υπόψη με την ε, διαδικασία της επιτήρησης και ότι οι δείκτες θα πρέπει να προσδιοριστούν και να ακολουθούν την πορεία του έργου να δίνουν ενημέρωση, feedback συγκεκριμένη για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος και να συλλέγονται όλα αυτά τα στοιχεία ταχύτερα. Είναι ζήτημα όχι μόνο του προγράμματος και του έργου, είναι ζήτημα λογοδοσίας απέναντι σε εσάς, απέναντι στο κοινοβούλιο. Να, να μπορείτε να παρακολουθείτε όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα ότι λειτουργεί καλά το έργο. Κύριε Γερμπράντη, την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε στην ε, ομάδα περιβάλλοντος του Συμβουλίου για να παρουσιάσουμε την ίδια έκθεση και θα δούμε τι είδους ε, ενδιαφέρον εμφανίζεται από εκείνη την πλευρά. Δεν ε, είμαστε ακόμα στο επίπεδο του ΕΚΟΦΗΝ, αλλά είμαστε πάντα στη διάθεσή τους εφόσον χρειάζεται να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας. Ξέρετε ότι έχουμε αρκετές ε, εκθέσεις συζητήσει μαζί και σε επίπεδο της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Ε, είναι μια γενική τάση των κρατών μελών, όχι μόνο για τη χρηματοδότηση για το περιβάλλον, αλλά και στην περιφερειακή ανάπτυξη κτλ. Να έχουν στο δυνατόν πιο ασαφείς και ευρύς στόχους, αφηρημένους στόχους, που θα δίσταζα ακόμα και στόχους να τους ονομάσω, έτσι ώστε να μπορεί να εγγραφεί το κάθε πιθανό πρόγραμμα μέσα σε αυτούς. Έχουμε υπογραμμίσει και σε πολλές ευκαιρίες Δυστυχώ όμω, αυτή την επίκριση, δυστυχώ όμω ε, η απάντηση από το Συμβούλιο είναι ότι α, χρειαζόμαστε ευελιξία και αυτό σε ένα βαθμό το δέχομαι, αλλά δεν μπορεί αυτό να παβαίνει ει βάρο τη διατύπωση σαφών στόχων και άρα τη δυνατότητα δυνατότητας προσμέτρησης της λειτουργίας των έργων αυτών, εάν ήταν σύμφωνα με του στόχου η εκτέλεση. Πολλέ φορέ εμεί ερμηνεύουμε τους στόχους που θα έπρεπε να επιδιώκει ένα έργο υπό το φως των ε, γενικόλογων θέσεων που έχουν εκφράσει τα κρατη Και από την άλλη πολλές φορές λέμε ότι και η Επιτροπή έχει προφανώς το δικαίωμα να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με τα προγραμματικά έγγραφα στη μακρο ή, μικρο, ή μικροπρόθεσμη βράχη πρόθεσμη διαχείριση, άρα μπορεί και η Επιτροπή να επικρίνει τους στόχους και την, την επιδίωξη των στόχων από τα προγράμματα. Επίσης, το ελεγκτικό συνέδριο έχει μια παράδοση. Σε κάθε έκθεση εκτέλεσης συνεχίζουμε την παρακολούθηση για δύο με τρία χρόνια. Δηλαδή θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε, παρακολούθησε τις ε, συστάσεις και τις επικρίσεις μας σε σχέση με την εκτέλεση αυτή και θα ενημερώσουμε αντίστοιχα το Κοινοβούλιο. Όπως είπα, κάνουμε κάθε τι το δυνατό ώστε να έχουμε το ταχύτερο δυνατό έτοιμε στι εκθέσει μα για το Κοινοβούλιο. Να γίνεται σωστά ο δημοσιονομικό έλεγχο και να σα προσφέρουμε επαρκή και έγκαιρη βέβαια ε, συμπεράσματα για την εκτέλεση των έργων. Για την κυρία Βελιέ. Προτιμώ να αφήσω τις ε, απαντήσει στην Επιτροπή, στην οποία απευθύνονταν οι ερωτήσεις. Δεν θέλω να κάνω σχόλιο πολιτικού τύπου. Και για την κυρία Ρομπότσοβα, Λιμπότσοβα, με χαρά σημειώνω ότι εάν είναι ικανοποιημένα τα κράτη-μέλη, εμείς εδώ έχουμε καλύψει πέντε κράτη-μέλη, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνων που περισσότερο αξιοποιούν τα κονδύλια του προγράμματος LIFE. Δεν μπορούμε να δώσουμε βαθμούς καλύτερος μαθητής, δεύτερος μαθητής κτλ. Απλώς εμείς με το δείγμα που έχουμε από τα πέντε κράτη-μέλη μπορούμε, να... μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, αλλά ήταν αντιπροσωπευτικό το δείγμα. Μπορεί να μην είχε επιλεγεί στο δείγμα μας η Βουλγαρία, αλλά δεν νομίζω ότι θα είχαμε κάτι, κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα αν ήταν και εκείνη μέσα. Αυτά λοιπόν και δίνω το λόγο στη συνάδελφο για να καλύψει τα λοιπά θέματα. Σε ό,τι αφορά την αύξηση του κόστους και σε ό,τι αφορά αυτήν την ομάδα παρακολούθησης, το monitoring team, θέλω να σας πω απλά ότι αυτή η ομάδα είναι ήδη επιχειρησιακή, ουσιαστικά είναι μια κοινοπραξία που βοηθά την Κομισιόν στην παρακολούθηση και την εφαρμογή των εργασιών στο πλαίσιο των έργων, των projects. Εμείς το μόνο το οποίο είχαμε συστήσει είναι να βελτιωθούν ορισμένε πρακτικές, ιδίως ό,τι αφορά την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων. Δηλαδή να παρακολουθείτε εξονυχιστικά ότι φέρνουν σε πέρας ε, στο πλαίσιο των προγραμμάτων ε, οι επιχειρήσεις όλες αυτές τις δραστηριότητες που έχουν αναλάβει. Θέλαμε να δούμε ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος ε, των έργων, πώς επηρεάζουν οι δραστηριότητες διάδοσης, τέτοιου είδους πράγματα. Δεν ζητάμε δηλαδή αύξηση του κόστους, αύξηση των δαπανών, αλλά βελτίωση σε ό,τι αφορά την ε, δραστηριότητα αυτής της ομάδας. Τώρα, την ερώτηση για το κλίμα. Θεωρώ ότι είναι ερώτηση που απευθύνεται πιο πολύ προς την Κομισιόν είναι λίγο ο προπολογισμό πράγματι, οπότε ο βασικό στόχο θα είναι η διενέργεια μελετών και συντονισμός πιο πολύ άλλων δράσεων για να είναι πιο καλή η εφαρμογή των πολικών, αλλά δεν μιλάμε για μεγάλες δράσεις, γιατί πραγματικά, όπως είπατε, δεν υπάρχει επαρκής προπολογισμός για κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ για Χαουκ. Για τα δημοσιονομικά μέσα, είχα μια ερώτηση. Πώς αξιολογείται την αξιοποίηση, αυτό που είπε και η κυρία Μπελιέ, την αξιοποίηση των δημοσιονομικών μέσων για την πολιτική. Όταν δεν έχουμε αρκετά χρήματα στη θέση μας, δίνουμε στις τράπεζες τα κονδύλια αυτά για να τα εφαρμόσουν, για να τα υλοποιήσουν, να υλοποιήσουν μέσω αυτών και την κλιματική πολιτική. Θεωρείτε ότι είναι επαρκές το σύστημα αυτό, γιατί και στην έκθεση για το παλιό πρόγραμμα LIFE είχατε επισημάνει πολλές φορές ότι δεν ήταν εστιασμένη επαρκώς η αξιοποίηση των κονδυλίων. Με αυτά τα δημοσιονομικά λοιπόν μέσα τα καταφέρνουμε ή τι πρέπει εν πάση περιπτώσει να προσέξουμε, πού πρέπει να δώσουμε την έμφαση. ώστε να ε, εξασφαλίσουμε αυτή την εστίαση, τη συγκέντρωση των κονδυλίων στον επιδιωκόμενο στόχο. Sie? Well, I... Φοβούμαι ότι δεν είμαι σε θέση να σας πω αυτή τη στιγμή ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτών των ε, μέσων. Σίγουρα θα είναι λιγότεροι οι πιθανοί στόχοι στους οποίους ε, θα αφοσιωθεί το live. Γιατί στο προηγούμενο live υπήρχαν γύρω στις 12 βασικές προτεραιότητες ε, που κάλυπταν τα πάντα, σε όλο το φάσμα και με τις ε, ενδεικτικές εθνικές πιστώσεις υπήρχε ένα πολύ ευρύ φάσμα ε, έργων και εκεί υπήρχε το πρόβλημα και με τον ανταγωνισμό και δεν υπήρχε μια κρίσιμη μάζα επιτυχημένων ε, έργων. Θέλουμε όμως να υπάρχει κάποια αισθητή βελτίωση, κάποια αποτελέσματα στην περιβαλλοντική πολιτική. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό το μέσο είναι το πλέον κατάλληλο για τη στόχευση, για την εστίαση. Αν κατάλαβα βέβαια καλά και το ερώτημά σας, ο προγραμματισμός ε, και η σαφή στοχοθέτηση για το life, Αυτά είναι τα βασικά, αν κατάλαβα καλά. Δεν βλέπω να είστε κανείς άλλο στο λόγο, η Επιτροπή. Παρακαλώ, από τη Γενική Διεύθυνση για το Κλίμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα δώσω το λόγο σε συνάδελφό μου για το κλίμα και για το πολιετέ και δράσης, αλλά θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κίνστ που υπογράμμισε ότι το περιεχόμενο αυτό τη έκθεση ε, που μας καθοδήγησε επηρεάζει και το πολιετέ πλαίσιο, ε, αλλά και τι προκήρυξει διαγωνισμών που θα ακολουθήσουν. Να πω το εξή. Πρώτα απ' όλα, κάποια από τα έργα που επισημαίνει και σχολιάζει το Ελληνικό συνέδριο χρηματοδοτήθηκαν ε, στο προηγούμενο, ε, στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος ε, που ήταν λιγότερο ξεκάθαρο το πεδίο εφαρμογή σε σχέση με το Life Plus. Και είχαμε τους δείκτες τώρα που είναι υποχρεωτικοί στο Life Plus για την απόδοση, για το output, αλλά δεν υπήρχαν πριν. Οπότε υπήρχαν κάποιες λήψεις στο προηγούμενο πρόγραμμα Life σχέση με τους δίκτες. Δεύτερο, η συμπατριώτησά μου ανέφερε κάποια ζητήματα αν αυτό το μικρό πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτήσει την ε, ε, διόρθωση ε, στην απώλεια βιοπικιλότητας και την αποκατάσταση για τις οδηγίες, για τα ενδιαιτήματα των ατόρων είναι ξεκάθαρα νομίζω και πιστεύω ότι τα ποσά στο πλαίσιο αυτής της αποκατάστασης βιοπικιλότητας και των συναφών δικτών Σίγουρα είναι πολύ λιγότερες, ε, μάλλον είναι πολύ ψηλότερες οι φιλοδοξίες μας, αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συλλέξουμε πόρους χρήσιμους για την ανάπτυξη πέτρου και από το Ταμείο Συνοχής και θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους αυτούς, αν βέβαια συμφωνούμε με τη συγκεκριμένη αυτή νομική βάση για τις ε, πτυχές του Νατούρα και της ε, βιοπικιλότητας, θα μπορούσαμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για την αποκατάσταση από όλες τις βιοπικιλότητες συνάδελφος. Για το υποπρόγραμμα κλίμα, στο νέο πρόγραμμα LIFE, αν δείτε τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στον τομέα του κλίματος, έχουμε τρεις στόχους για το 2020. Για τα θερμοκηπιακά αέρια, τις εκπομπές, εδώ είμαστε στο στόχο μας. Θέλαμε να έχουμε μέχρι το 2020 20% έμπω στο 18% για τις ανανόσιμες πηγές και εδώ πιστεύω θα φτάσουμε το στόχο μας και υπάρχει και ένας τρίτος στόχος που είναι η ενεργειακή απόδοση. Αλλά εδώ απέχουμε πόρο του να είμαστε στη σωστή κατεύθυνση και για να πετύχουμε το στόχο αυτό χρειάζονται ειδικά μέσα και εργαλεία, να έχουμε δηλαδή μεγαλύτερη χρηματοδότηση για μέτρα ενεργειακή απόδοση. Θέλουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή με το πρόγραμμα LIFE. Ο τομέα αυτό ε, ε, νομίζω ότι μπορεί να καλυφθεί με το LIFE, ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση. Τα σχετικά έργα έχουν το πρόγραμμα ότι θα είναι ε, προγράμματα που θα βοηθήσουν στη μείωση του κόστους, εξοικονόμηση θα έπρεπε να πω ότι οι επιδοτήσεις είναι ένας δαπανηρός τρόπος χρήσης των δημοσίων ε, κονδυλίων. Βέβαια, ο ιδιωτικός τομέα ή μάλλον ο χρηματοοικονομικό τομέα, τα δάνεια αυτά λόγω διαρθρωτικών προγραμμάτων δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει, ιδίω ο τραπεζικός τομέα. Δεν έχει αντιληφθεί αυτό το κομμάτι της αγοράς ότι υπάρχει και δεν συμμετέχει. Επίσης τα έσοδα είναι μικρά συνήθως. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ενδιαφέρον επιχειρηματικό αρκετό. Μπορούμε να δοκιμάσουμε και νέα ε, προγράμματα χρηματοδότησης στο τραπεζικού τομέα. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα συνεργαστούμε με τις τράπεζες των κρατών μελών που μπορούν άμεσα να, αποπληρω... να ε, δώσουν δάνεια σε... για μικρά έργα που αναλαμβάνουν ε, νοικοκυριά ή μικρές επιχειρήσεις για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Έχουμε 80 εκατομμύρια, δεν είναι και πολλά χρήματα, αλλά θα μπορέσουμε να δοκιμάσουμε αυτό το ε, πρόγραμμα σε κάποια κρατημέλη και μετά από λίγα χρόνια θα γνωρίζουμε πώς λειτουργεί. Ήδη είδαμε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει αυτή η επανάληψη, αντιγραφή προγραμμάτων μέσω των διαθετικών ταμείων. Άρα υπάρχει ε, μεγάλη πιθανότητα να μπορέσει αυτό το νέο μέσο που δοκιμάζεται και είναι ένα κεντρικά διαχειριζόμενο έργο, να μπορέσει να επαναληφθεί από τις περιφέρειες, από τα κράτη-μέλη μέσω των διαθετικών ταμείων. Δυνητικά λοιπόν θα είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αξιοποίησης των δημοσίων κονδυλίων. Ταυτόχρονα έχει πολύ μεγάλη σχέση και με τις εθνικές πολιτικές για την ενεργειακή απόδοση. Το εργαλείο αυτό, το, ο μηχανισμός αυτός θα, θα συνδέεται με αυτό το σχέδιο δράσης που θα πρέπει να εγκρίνουν μέχρι φέτος τον Απρίλιο όλα τα κράτη-μέλη. Άρα για να είναι επιλέξιμο ένα έργο για χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι επιλέξιμο και για αυτά τα εθνικά προγράμματα. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένα πρόγραμμα σε ένα κράτος μέλος όπου έχουμε 5% επιδότηση στις έργα ενεργειακής απόδοσης. Ωστόσο, η επιχείρηση, των νοικοκυριό, τι θα γίνει, πώς θα μπορέσει να αποκτήσει αυτό το 95% το υπόλοιπο ε, της χρηματοδότησης. Θα μπορούσε εδώ να υπάρξει ένα συνδυασμός εθνικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Είναι μια καλή ευκαιρία να δοκιμάσουμε ένα νέο μηχανισμό, ένα νέο εργαλείο. Ένα άλλο εργαλείο που θα δοκιμάσουμε είναι μια, ένα άλλο εθνικό μέσο, μια πιλωτική φάση για να δούμε τη νέα χρηματοδότηση, παραδείγματο χάρη προσαρμογή στι κλιματικέ αλλαγέ. Ξέρουμε ότι είναι τεράστιο το κόστο για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών που παρατηρούμε στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε επίση ότι τα, οι δημόσιοι πόροι δεν θα αρκέσουν για την αντιμετώπιση τη πρόκληση αυτή. Υπάρχει λοιπόν έντονη ανάγκη να δοκιμάσουμε, να δούμε πώ μπορούμε ε, να εμπλέξουμε και τον ιδιωτικό τομέα στη χρηματοδότηση. Έχουμε λοιπόν αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που θα δει διάφορου τρόπου ε, με του οποίου θα μπορούσε να συμμετάσχει ο ιδιωτικό τομέα στη χρηματοδότηση. Προτείνουμε λοιπόν ε, δύο χρηματοδοτικά μέσα, αυτά τα δύο που σα προανέφερε, να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα LIFE. Ευχαριστώ. Να πηγαίνατε και στο συλλογικό όργανο της Επιτροπής, να τους πείτε τα ίδια πράγματα και να σας ακούγανε και εκείνοι. Το 2000, για το 2030 έχει ορίσει στόχους το Κοινοβούλιο, αλλά η Επιτροπή δεν είχε το θάρρος και το ανάστημα για να τους ορίσει, για να ορίσει συγκεκριμένες προτάσεις ε, στα θέματα της των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έμεινε υπερβολικά σαφής γιατί δεν τόλμησε, αλλά εν πάση περιπτώσει και ευτυχώς τελειώνει η θητεία αυτής τη Επιτροπής και έρχεται μια καινούρια και ελπίζουμε ότι αυτοί θα είναι σε θέση 100% να αγωνιστούν για αυτού του στόχου. Όπω του παρουσιάσατε άλλωστε και εσεί και ελπίζω να με ακούει κάποιος από τι σχετικέ υπηρεσίε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μόλι μα παρουσιάσατε. Έτερο θέλει το λόγο. Όχι, ε, τότε ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνιστώ να συζητήσετε και εσωτερικά στις υπηρεσίες σας αυτές τις θέσεις. Κύριε Κίνηση, θα έχετε κάτι να συμπληρώσετε. Καταρχάς και πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όπως είπα την περασμένη φορά που εξετάσαμε το πρόγραμμα LIFE και τις νέες προκλήσεις που αυτή τη στιγμή καλύπτονται στον κανονισμό, ε, να πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον να εξετάσουμε το πρόγραμμα αυτό και τα αποτελέσματά του. Θα επαναλάβω κάτι που είπα και στην αρχή. Εάν στον νέο κανονισμό υπάρχει κάτι που θα έπρεπε να λύεται με τα εξασιοδότηση πράξης είναι η παράγραφος στο εδάφιο 3 με το σημείο 3, δηλαδή οι δείκτες των επιδόσεων. Αυτοί οι δείκτες, όπως αναφέρονται εδώ, θα πρέπει να, να είναι αντικείμενο καλύτερης επεξεργασίας και τονίζουμε στην εκθεσή μας ότι οι γενικοί προσανατολισμοί των δικτών επιδόσεων θα πρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο στα αποτελέσματα με κάποια ερωτηματικά διότι οι δείκτες επιδόσεων, λόγω χάρη ο αριθμός παρεμβάσεων που εφαρμόζονται αναστατηγική πρόγραμμα ή ο αριθμός παρεμβάσεων που είναι επιλέξιμες για την χρηματοδότηση ή τη μεταφορά. Αυτός ο σχεδιασμός δικτών έχει να κάνει περισσότερο με με την παραγωγή ε, και όχι τόσο με τα αποτελέσματα ή με τα επιτεύγματα. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίζει τις της πράξεις ανάλογα με τις με τις προοπτικές των δικαιούχων και είναι απαραίτητο νομίζω σε αυτό το σημείο. Κατά τα άλλα, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για τον ενδιαφέρον που έδειξε για την εκθεσή μας και σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κίντς. Έγινε πολύ καλή συζήτηση, ελπίζω με μεγάλη προσοχή να παρακολούθησαν όλοι, τα θεσμικά όργανα δηλαδή, τα όσα υπόθηκαν. Ολοκληρώνουμε το θέμα αυτό της ημερησίας διάταξης, το υπαριθμόν 4 και προχωρούμε ως εκ τούτου με τον Καρλ Σλίτερ και την ένστασή του. Uh, Ευχαριστώ. Θα μείνετε εδώ. Καλά. διάβασα τον κατάλογο των κατεξουσιοδότηση πράξεων και είδα κάτι για τη μεταφορά των ε, λοιπόν στη θάλασσα και των ελαίων. Δεν μου άρεσε. Εάν θέλει κανείς να μεταφέρει βρόσιμα έλαια, θα πρέπει να έχει ειδική δεξαμενή. Έπειτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ε, εξήγησε ότι είναι δύσκολο, δημιουργεί προβλήματα, είναι δαπανηρό, να κάνουμε αυτό που κάνει βάσει των καταφεντηρίων γραμμών της η βιομηχανία, δηλαδή οι εταιρείε πέραν των πλέον επικίνδυνων χημικών που δεν μπορούν να βρίσκονται στο προηγούμενο φορτίο. Ε, αναλύθηκε αυτό και από την ΕΦΣΑ και είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αρκεί να καθαρίζονται δεξαμενέ. Εάν δείτε όμω κάποιε από τις ουσίες ακόμη και βάσει των προτύπων του βιομηχανικού κλάδου μερικά είναι επικίνδυνα, όπως τα λευκά μεταλλικά έλαια, μεταλούχα έλαια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν προβλέπει καν αυτήν την ε, απέτηση, διότι ακόμη και μια μικρή περίπτωση ύπαρξη των ε, ουσιών αυτών υπάρχει, όπως οι ουσίες CM2, που είναι ιδιαίτερα τοξικές, τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ δύσκολα. Για την ΕΦΣΑ λοιπόν αρκεί ο καθαρισμός των δεξαμενών. Εγώ δεν είδα πουθενά καμία απέτηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους ε, υπευθύνους να ελέγχουν την καθαριότητα των δεξαμενών. Πώς ξέρουμε ότι καθάρισαν τις δεξαμενές σε κάθε περίπτωση. Και για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι για να συμμορφωθεί κανείς με την απέτηση της ΕΦΣΑ να είναι καθαρές οι δεξαμενές, λόγου χάρια. Για ένα από τα κοινά πρόσθετα του, α, της βενζίνης. Είναι πολύ κακή η γεύση του όταν μεταδοθεί στα τρόφιμα, ο μεθυλεθέρας και είναι ένα επικίνδυνο χημικό. Τι γίνεται αν χρησιμοποιηθεί αυτό το πλοίο και καθαρίσουμε τις δεξαμενές και τελικά καταλήξει στο νερό ε, της Ευρωπαϊκής, στο υδροδοτικό σύστημα. Τι μέτρα υπάρχουν για την προστασία του περιβάλλοντος, αν χρειαστεί. Και υπάρχουν και άλλες ουσίες τις οποίες βρίσκω περίεργες και δεν βλέπω να υπάρχουν διασφαλίσεις ότι οι απαιτήσει της ΕΦΣΑ να είναι καθαρές δεξαμενές θα εφαρμόζονται. Πέραν όλων αυτών, νομίζω οι περισσότεροι Ευρωπαίοι τι θα σκεφτούν. Μισό λεπτό, ακόμα και αν δεν είναι ε, επικίνδυνο, είναι πολύ περίεργο να έχει περάσει το δικό μου το λάδι που χρησιμοποιώ στην κουζίνα μου από μια δεξαμενή με θήκο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα ήθελα να μου το εξηγήσει. Υπάρχει σίγουρα στρατηγική καθαρισμού και ελέγχου του καθαρισμού των δεξαμενών. Ιδάλλως ε, εμένω στην αστασή μου κατά της πρότασης αυτής. Καλώς. Και παρακαλώ την Επιτροπή να λάβει το λόγο. Αυτό το λόγο κύριε Βουλή. Σε... Ευχαριστώ πρόεδρε. Το σχέδιο αυτό κανονισμού είναι μια προσαρμογή της νομοθεσίας που υπάρχει από το 1996, δηλαδή πάνω από 18 χρόνια. Συστηματικά επικαιροποιούμε τον κατάλογο των χημικών ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις δεξαμενές των πλοίων και μπορεί να υπάρξουν εκεί πριν τη μεταφορά ελαιόλαδου. Ελαίων για την ανθρώπινη κατανάλωση, βρόσιμων υγρών ελαίων δηλαδή. Έχουμε πέντε επιχειρήματα για να προσπαθούμε τη θέση μας. Πρώτον, ότι εδώ και 18 χρόνια που υπάρχει και εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία, η κοινοτική νομοθεσία αποτελεί πρότυπο για τις τρίτες χώρες, ιδίως για τις αναπτυσσόμενες, από τις οποίες εισάγουμε αυτά τα λύπη. Οι ίδιοι δεν έχουν την κατάλληλη νομοθεσία, τις επιστημονικές γνώσεις για να μπορέσουν να εκπονήσουν τη σχετική νομοθεσία. Εργαζόμαστε συστηματικά σε επίπεδο κόντεξ, ε, ώστε ο κατάλογος των ε, χημικών ουσιών που μπορούν να εγκρίνονται και να επιτρέπονται επικαιροποιείται. Αυτό είναι μια σημαντική προσπάθεια, διότι θέλουμε να είναι πλήρης ο κατάλογος των χημικών ουσιών. Και ακριβώς γιατί δεν θέλουμε να υπάρχει και μεταφορά επικίνδυνων χημικών ουσιών. Το δεύτερο επιχείρημα είναι οικονομικής ε, διάσταση διότι τα σκάφη αυτά που μεταφέρουν τα έλαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να φύγουν άδεια. Ένα πλοίο δεν πλέει στη θάλασσα κενό. Αυτό είναι αδύνατο. Πρέπει λοιπόν να ξαναφύγουν με κάτι, κάποιο περιεχόμενο στις δεξαμενές τους. Εάν έφευγαν κενά, οι οικονομικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο κόστος ε, της εισαγωγής ελαίων ή λοιπόν για διάφορες χρήσεις, είτε για την ε, εκτροφή των ζώων είτε για την ανθρώπινη κατανάλωση, θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 6%. Και το τρίτο επιχείρημα έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος. Τα σκάφη αυτά, όπω είπα, δεν μπορούν να φεύγουν άδεια. Εάν δεν υπάρχει κάποιο περιεχόμενο ή κάποιο προϊόν στις δεξαμενές, πρέπει για να υπάρχει σωστό έρμα να ε, έχουν θαλασσινό νερό στις δεξαμενές. Όμως το πρόβλημα είναι ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει περιβαλλοντικές επιπτώσεις η μεταφορά του νερού. Μπορεί να μεταφερθεί φυτοπλανκτόν που να είναι τοξικό λόγου χάρη. Έτσι εισήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τοξικά φυτοπλανκτών που προκαλούν την, ε, ε, για τα δίθυρα μαλάκια, ε, δηλαδή τα στρίβια, τα μύδια και άλλα όστρακα, την τοξική παράλυση. Και αυτά ήρθαν ακριβώς από το νερό που χρησιμοποιεί το σέρμα. Έπειτα, δεν έχουμε περιστατικά μόλυνσης είτε από τοξικές ουσίες είτε από αποβάθμιση της ποιότητας των ε, ελαιών. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν καταγράφει από τις Εθνικές Αρχές την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και 18 χρόνια που η πρώτη νομοθεσία εγκρίθη, ενεκρίθη από το 1996 δηλαδή. Θα σας φαίνεται περίεργο, σίγουρα, το θικό να μεταφέρεται σε μια πρώτη φάση στην ίδια δεξαμενή που μετά θα καθαριστεί και θα μεταφέρει γραέλαια. Είναι κάπως περίεργο. Όμως αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε πρόσφατα από την ΕΦΣΑ να επαναξιολογήσει περίπου μια εκατοστή χημικές ουσίες που βρίσκονται σε, αυτήν, σε αυτόν τον κατάλογο εδώ και 18 χρόνια και αυτό είναι το πέμπτο με επιχείρημα, αξιολόγησε όλες τις ουσίες η ΕΦΣΑ. Απορρίφθηκαν πέντε, τις οποίες τις εξαλείψαμε από τον περιβόητο κατάλογο, το περιβόητο αυτό παράρτημα. Όμως, η ΕΦΣΑ θεώρησε τις τρεις ουσίες για τις οποίες μιλά ο κύριος Σλίτερ στην ε, πρότασή του, στην πρόταση ψηφίσματος, αυτές τις αξιολόγησε θετικά. Το περίφημο MTBE το οποίο κατά τον κύριο Σλίτερ προκαλεί ζαλάδες ε, λόγω της οσμής του από την τότε Επιστημονική Επιτροπή το 1996 θεωρήθηκε ε, μετά από τρεις επιστημονικές αξιολογήσεις και εφόσον οι δεξαμενές του πλοίου καθαριστούν, θεωρήθηκε ότι δεν παρουσιάζει πρόβλημα. Για τα λευκά ορυκτά έλαια θεωρήθηκε ότι αυτά δεν προορίζονται άμεσα για την ανθρώπινη κατανάλωση, οπότε δεν υπάρχει σχετικός κίνδυνος και προτείναμε ακριβώ αυτό το παράρτημα που καταργεί πέντε ουσίες οι οποίες ήδη περιλαμβάνονταν στον κατάλογο. Το παράρτημα αυτό το στηρίξαμε με πολύ με αναντήρητα και ελεγμένα επιστημονικά στοιχεία και τώρα για, το, για την πλήση των ε, δεξαμενών του πλοίου πριν την φόρτωση υγρών ελαίων. Ο καθαρισμός αυτός γίνεται σε τρίτες χώρες αφού αδειάσουν οι δεξαμενές από χημικές ουσίες και τότε φορτώνονται τα υγρά ελαία. Δυστυχώς δεν έχουμε νομικό τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις τρίτες χώρες που ε, μας δίνουν τα ελαιά τους, δεν έχουμε την δυνατότητα να επιβάλλουμε υποχρεώσεις από νομική σκοπιά. Γι' αυτό το λόγο στην νομοθεσία μας προβλέπεται ο καπετάνιος του πλοίου, ο, κυβερνήτης, που είναι υπεύθυνο για τα προϊόντα που μεταφέρονται, ε, να παρέχει όλες τις γραπτές εγγυήσει στον ευρωπαϊκό λιμένα όπου προσαράζει το σκάφος και οι υγειονομικοί ελεγκτές κάνουν τον ελεγχό του. Πρέπει λοιπόν να παράσχει όλες τις ε, γραπτές εγγυήσει ότι ο καθαρισμός έγινε βάσει των διεθνών κανόνων. Υπάρχουν διεθνεί κανόνες για το θέμα αυτό και συγκεκριμένα ότι δεν έγινε η πλήση ε, στα ανοιχτά, στη θάλασσα και ότι τα νερά αυτά δεν ε, έπεσαν μετά στην θάλασσα. Αυτά τα νερά πρέπει να συλλέγονται και να διατίθενται προκειμένου να αποφευθεί η, η της θάλασσας ή των λιμένων που, ε, όπου προσαράζουν τα σκάφη. Ιδού, Πρόεδρε, τα νομικά και οικονομικά επιχειρήματα που μας έκαναν να υποβάλουμε αυτή την πρόταση κανονισμού. Σας ευχαριστώ. Vielen Dank. Gibt es weitere Θέλει κανείς λόγο. Very briefly. Uh, πολύ σύντομα. Υπάρχουν κίνδυνοι. Υπάρχουν όμως τελικά. Γιατί λέει η Κομισιόν δεν υπάρχουν. Και γι' αυτό στρέφομαι σε σένα, Κάρλ, γιατί κατέθεσα αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ένσταση και σε ρωτώ. Εσύ αυτό που μας είπε η Κομισιόν ε, μπορείς να το διαψεύσεις, ε, γιατί μένα με πείθουν αυτά που άκουσα από την Κομισιόν. Ο Καρλ Λιούτερ. Ακούστε, για κάποιες ουσίες συμφωνώ με την Κομισιόν ότι δεν αποτελούν κίνδυνο, γιατί υπάρχουν κάποιες ε, ουσίες που δεν είναι επικίνδυνες και ακόμη και αν δεν καθαριστεί η δεξαμενή και παραμείνουν σε υπολείμματα, αυτής δεν θα είναι καταστροφικό. Ε, ακόμη και αν ε, ακούγεται έτσι πολύ άσχημο το θήκο οξύ, επειδή θα διαλυθεί και θα είναι πάρα πολύ μικρή περιεκτικότητά του μέσα στο υγρό που θα μπει, ίσως να μην είναι τόσο πολύ επιβλαβές, αλλά για το MTB, τον μεθυλοτριτό βουτιλεσθέρα, ε, 15 μικρογραμμάρια του λίτρου ε, θα μπορούσε να είναι υπερεκτικότητα και εκεί είναι επικίνδυνο. Άμα διαβάσετε γνωμοδοτήσει τη ΕΦΣΑ και έχω διαβάσει εγώ τέτοιε γνωμοδοτήσει, πάντα εκεί θεωρούν ω υπόθεση παίρνουν ε, ότι είναι καθαρέ οι δεξαμενέ. Η Κομισιόν όμω επισήμανε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα τουλάχιστον από μικρή πλευρά να το επιβεβαιώσουμε αυτό, για το τι συμβαίνει στι τρίτε χώρε. Δεν έχουμε εγγυήσει δηλαδή ότι μπορεί, μπορεί να μην ε, είναι καθαρέ οι δεξαμενέ. Και στη σύμβαση του Χονγκ Κονγκ. Δύσκολο να ρυθμιστούν οι διεθνεί ε, ε, ναυτιλιακές μεταφορές. Για 15 χρόνια παραβιάζονταν οι όροι και δεν το καταλάβαινε κανείς και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η Κομισιόν λέει, α, δεν υπάρχει πρόβλημα, καθαρίζονται παντού οι σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Το θέμα είναι αν το πιστεύει κανείς ή όχι, γιατί ναι, αν τις καθαρίζουν, φυσικά συμφωνώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι ασφαλής. Αμφιβάλλω όμως ότι είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αυτό και δεν ξέρω και κατά πόσο θα το πιστέψουν και οι καταναλωτέ. Δηλαδή δεν διαφωνώ με, το, με την Κομισιόν επί δηλαδή ότι αν η δεξαμενή είναι καθαρή, ασφαλή. Συμφωνώ. Συμφωνώ από αυτού. Η ένστασή μου βασίζεται στο ότι δεν έχουμε νομικά μέσα στη διαθέσή μα για να επαληθεύσουμε ότι καθαρίζονται δεξαμενέ. Ούτε και από διοικητική πλευρά μπορούμε να το διασφαλίσουμε αυτό. Εκεί έγκυται η διαφωνία μου και όχι στα επιστημονικά στοιχεία το θέμα είναι ότι έχουμε εκεί μεγάλο κίνδυνο να μην είναι τα πράγματα όπως θέλουμε να είναι, να μην καθαρίζονται δηλαδή δεξαμενές. Και εξακολουθώ να διαρωτώ με, γιατί δεν ζήτησε η Κομισιόν. Γιατί για να σας πω και έτσι να είμαστε και ειλικρινείς, αυτός ο κατάλογος είναι αντιγραφή από τον κατάλογο των επιχειρήσεων. Όμως επιχειρήσεις ζητάνε και έχουν κάποιες απαιτήσεις και για το ρηκτέλεα. Ε, τα λευκά ορικτέλα. Μπορεί να έχουν κάποια καρκινογόνα επίπτωση, δεν ξέρω. Γιατί δεν τα πήρατε όλα αυτά που ζητάει ο κλάδος των επιχειρήσεων και μόνο, τον, ε, μόνο αυτή τη λίστα. Γιατί στα ορυκτέλα τα λευκά νομίζω ότι το παραφινέλο πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Μήπως πρέπει εδώ να πούμε τι είδους διαστάσεις, ε, όγκοι, καλύτερα ποσότητες αναφέρονται εδώ. Αυτό ζήτησε ο κύριος Λίτερ. Παρακαλώ η Επιτροπή. Πρόεδρε, δεν είμαι ακριβώ σε θέση να απαντήσω στην ερώτησή σα. Όμω οι ποσότητε που μεταφέρονται ένα σκάφο μπορούν να φτάσουν τα 500 λίτρα. Όχι, 100 κυβικά μέτρα. Μιλάμε για ποσότητες ε, μεγάλες που χρησιμοποιούνται είτε για την ε, τροφή των ζώων, για τη ζωική κατανάλωση, δηλαδή εκεί κατευθύνονται, για τους χείρους της ε, Αγελάδες, τα βοηθεί και τα πτηνά, τις όρνηθες και όχι για την ανθρώπινη τόσο πολύ. Αλλά να απαντήσω στον κύριο Σλίτερ. Δεν υποτιμούμε τον κίνδυνο. Απλώς προσπαθούμε να τον ελαχιστοποιήσουμε διότι ακριβώς ελέγχουμε τον κατάλογο των χημικών ουσιών. Δεν επιτρέπονται όλες, 100 είναι χημικέ ουσίε που αναφέρονται εδώ ε, είναι αρκετά σοβαρό αριθμό σε σχέση με το σύνολο των χημικών ουσιών που μπορούν να μεταφέρονται από πλοίο. Τώρα για το πρόβλημα τη πλήση των δεξαμενών. Πρέπει να υπάρχει ε, γραπτή έγκριση από τον κυβερνήτη του πλοίου, διότι πιστεύουμε χωρίς να θέλουμε να κρίνουμε τις δυνατότητες των αρχών στις τρίτες χώρες, είναι διεθνής κανόνας. Ο κυβερνήτης του πλοίου είναι υπεύθυνος για το φορτίο που μεταφέρει. Γι' αυτό λοιπόν προτιμούμε να ισχύει η γραπτή έγκριση η οποία περνάει από τον έλεγχο των τελωνιακών και υγειονομικών αρχών όπου προσαράζει το πλοίο στην άφηξη και έπειτα μην ξεχνάμε τους ελέγχους κατά την άφηξη ακριβώς είναι στο συμφέρον των εταιρεών που αγοράζουν αυτά τα υγρά, έλαια, η λύπη, είτε για ανθρώπινη είτε για ζωή και κατανάλωση, τα λύπη αυτά ακριβώ να μην έχουν μολυνθεί με ουσίε που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην ε, ζωή και την ανθρώπινη υγεία. Όπω είπε ο κύριο Σλίτερ, το MTB είναι μία ουσία που προκαλεί δυσοσμίε. Αμέσω ανοιχνεύεται λοιπόν, εάν οι δεξαμενέ δεν είναι καθαρισμένες, εάν υπάρχουν κατάλοιπα, σε ποσότητα μεγαλύτερη των 100 mg ανά κιλό, τότε οι οσμές αυτές δείχνουν ότι η πλήση δεν έγινε σωστά. Το φορτίο λοιπόν απορρίπτεται. Δεν γίνεται δεκτό μάλλον. Το επαναλαμβάνω, εδώ και 18 χρόνια που ισχύει η νομοθεσία αυτή, δεν υπήρξε κανένα περιστατικό ή ατύχημα, δεν κατεγράφει τίποτα από τα κράτη-μέλη, ούτε από τις εταιρείες του βιομηχανικού κλάδου. Okay, vielen Okay, Well, you Κοιτάξτε, συνεχίζετε να αποφεύγετε την ερώτησή μου για τα λευκά ορυκτέλεια. Και έπειτα, ακούσατε για το Έρικα, θυμάστε αυτό το ναυάγιο. Τα κάνετε να ακούγονται τόσο ε, απλά, φταίει ο κανένας. Για το Έρικα δεν υπήρχαν ευθύνες. 50 διαφορετικές εταιρείες ε, είχαν εμπλοκεί και κανείς δεν μπορούσε να ε, αναλάβει ευθύνη γιατί ο ένας κατηγορούσε τον άλλο. Και τότε καταρτίστηκε ότι μία εταιρεία ήταν υπεύθυνη για το φορτίο, μία άλλη για τη φόρτωση του φορτίου στο συγκεκριμένο πλοίο, μία άλλη για τη μεταφορά του. Υπήρχε ένα πλήρωμα με άλλη εταιρεία, μία ε, εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για τον κυβερνήτη και μία άλλη εταιρεία που ήταν η διοκτήτρια όλων των υπολείπων. Λοιπόν, ήταν πολύ δύσκολο να αποδοθεί ευθύνη. Και τρίτον, γιατί λέτε ότι θα μεταφερθεί θαλασσινό νερό. Αυτό είναι ανόητο. Αν φτάσει κανείς στο Γκέτεμπεργκ με άδειο, με σε ένα άδειο σκάφος, προφανώς θα εξάγει πόσιμο νερό. Γλυκό νερό δηλαδή. Στη Νομίζω ότι εδώ ξεχνάμε ανάπτυξη που μπορεί να έχουμε με αυτή τη δυνατότητα και θέσει απασχόληση στην Ευρώπη και όχι με ανοησίε περί μεταφορά θαλασσινού νερού. Θέλει η Επιτροπή να απαντήσει σε αυτό, κύριε Πουλή. Πράγματι, κύριε Πρόεδρε, δεν απήντησα στον κύριο Σλίτερ για τα εδόδημα. Έλα. Α, δεν υπάρχει λόγος να μην μεταφέρονται αυτά. Εδόδημα είναι δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν στην εξαίρεση. Η εξαίρεση και το παράτημα αφορούν τις ουσίες που δεν πρόκειται, δεν κατευθυνόνται στην κατανάλωση. Τα άλλα λευκά ορυκτέλεα που δεν προορίζονται για ανθρώπινη, για ζωική κατανάλωση. Η Εύσα μας είπε ότι αυτά τα λευκά ορυκτελεα εφόσον γίνει η πλήση και το δέχομαι ότι εδώ πρέπει να γίνει κάποια επιπλέον επαλήθευση. Αλλά εφόσον καθαριστούν οι δεξαμενέ του σκάφου, τα λευκά ορυκτέλεια μπορούν να μεταφέρονται πριν την πλήση και μετά να μεταφερθούν τα ε, δόδημα έλαια. Ναι, με το έρικα έγινε ναυάγιο και υπήρχε και ρήπανση των, ε, της ακτογραμμής με την πετρελοκυλίδα. Σαφώς. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για ατυχήματα, μιλάμε για έλεγχο της πιστοποίησης και των εγγράφων που υποβάλλει ο κυβερνήτης για να δούμε αν πλήθησαν, σωστά οι δεξαμενές του πλοίου. Τώρα τι να σας πω, μπορούμε να τον πιστεύουμε ή όχι, μπορεί να υπάρχουν ψευδοί ή όχι πιστοποιητικά. Ε, εάν ζητήσουμε από τις λιμενικές αρχές προέλευσης την ε, ε, πιστοποίηση ότι πλήθη σωστά ή όχι το σκάφος, και πάλι μπορεί να υπάρξει νοθεία η παραποίηση ενός πιστοποιητικού, αλλά βάσει των διεθνών κανόνων εμπορίου ξέρουμε ότι η πιστοποίηση από τον κυβερνήτη η πιστοποίηση της πλήσης των δεξαμενών για τη μεταφορά μετά εδόδημων ελαίων τηρουμένων των αναλογιών είναι ακριβώ η εγγύηση που απαιτείται. Ελπίζω ότι απέντησα στον κύριο Σλίτερ. Σας ευχαριστώ. Και έτσι τελειώνουμε τη συζήτηση. 19 Μαρτίου ψηφίζουμε. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει η ψηφοφορία τον Απρίλιο στην πρώτη σύνοδο. Και συνεχίζω πάλι με τον Καρλ Σπλίτσαρ και το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης Διεθνή Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ για την ασφαλική περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση των πλοίων 2009. Κύριε Σιγητά. Είναι η μέρα μου σήμερα. Θα θυμάστε. Σχόλιο του πρόεδρου μικροφώνα. Ε, μικροφώνου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα θυμάστε όταν συστήσαμε τον κανονισμό για την υλοποίηση της σύμβασης του Hong Kong στην Ευρώπη. Δική μου έκθεση. Η σύμβαση αυτή ορίζει διεθνή πρότυπα για τον παροπλισμό, τη διάλυση πλοίων. Τα πρότυπα αυτά όμως, κατ' με, αλλά και σύμφωνα με τους περισσότερους Ευρωπαίους, είναι πολύ χαμηλά. Θα θέλαμε να βελτιωθεί λοιπόν το σχετικό πρότυπο. Θα θυμάστε επίση ότι είχαμε και τη σύμβαση της Βασιλείας που απαγορεύει την εξαγωγή τοξικών αποβλήτων. Και καταρχήν όλα τα πλοία του μεγέθους που καλύπτει η σήμανση του Hong Kong μεταφέρουν τοξικά έλαια, τοξικές μπογιές, τοξικά χημικά, ηλεκτρολογικά κτλ. Έχουν PCB, έχουν αμίαντο πολλές φορές. Άρα πολλά από αυτά τα πλοία είναι γεμάτα από τοξικές ουσίες. Το πρόβλημα για τη βιομηχανία ε, ή μάλλον μπορεί να αποφύγει την ε, σύμβαση της Βασιλείας λέει ότι δεν μεταφέρει απόβλητα. Όταν φύγει όμως από τα ευρωπαϊκά ε, ύδατα λέει ναι, έχει τοξικά και θα το δούμε όταν φτάσουμε στην Ινδία. Και αυτό συμβαίνει στο 90% των περιπτώσεων. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες που θεσπίσαμε λόγω της πλήρους αποτυχίας εφαρμογής ε, της Σύμβασης της Βασιλείας δίνουν τη δυνατότητα, λοιπόν, επιτρέπουν την εξαγωγή αυτών των πλοίων ε, αποβλήτων, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρέ ε, προϋποθέσεις που τελικά όμως δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Ποιε είναι αυτές οι αυστηρέ προϋποθέσεις, περιλαμβάνουν αυτές τις κλές επιφάνειες, ε, τον εξοπλισμό για την διάλυση, τον παροπλισμό, την επεξεργασία των ανακτηθέντων αποβλήτων, περιλαμβάνουν διατάξεις για την προφύλαξη, την προστασία των εργαζομένων και ανακύκλωση των τοξικών ουσιών. Ουσιαστικά υπάρχουν λοιπόν προϋποθέσεις ε, που θα θέλαμε να ισχύουν και στην Ευρώπη. Ακόμη και αν κάποιος ε, εξάγει εντό αγωγικών προς διάλυση το πλοίο του σε μια άλλη χώρα. Εγώ θα συνιστούσα να ψηφίσουμε υπέρ της επικύρωσης της Σύμβασης του Χονγκ Κόνγκ, όμως η Σύμβαση του Χονγκ Κόνγκ δεν σημαίνει ότι θα εφαρμοστεί άμεσα. Μία μόνο χώρα, η Νορβηγία, έχει επικυρώσει μέχρι τώρα. Φαντάζομαι ότι επειδή δεν είναι μέλος της Ένωσης, είχε πιο πολύ χρόνο να ασχοληθεί με αυτό το θέμα και όχι με τα υγρά έλα για παράδειγμα. Αλλά τέλος πάντων, η Νορβηγία είναι η μόνη χώρα που μέχρι στιγμής έχει επικυρώσει τη Σύμβαση του Χονγκ Κόνγκ. Ο κανονισμός που εγκρίναμε θα τεθεί σε ισχύ το νωρίτερο την 31η Δεκεμβρίου 2015 και το αργότερο 31 Δεκεμβρίου 2018 ανάλογα με την δεσιμότητα και την ικανότητα για το πόσο θα γίνει αυτή, πώς θα εφαρμοστούν ε, οι διατάξεις. Αν εγκριθεί, μάλλον αν επικυρωθεί η σύμβαση του Χονγκ Κονγκ πριν τεθεί σε ισχύ ο δικός μας κανονισμός, θα υπάρχει ένα παραθυράκι ώστε να μπορούν να εξάγονται αυτά τα πλοία χωρίς να τηρούνται αυτές αυτέ τι προποθέσει. Αλλά δεν είναι τόσο πιθανό το σενάριο αυτό. Οι πιο πολλοί θεωρούν ότι η σύμβαση του Χονγκ Κόκ μάλλον δεν θα επικυρωθεί πριν το 2020. Και αυτό γιατί υπάρχουν πολλοί και διάφοροι όροι και προϋποθέσεις για το πόσε χώρε πρέπει να επικυρώσουν ε, πόσο ποσοστό της δυναμικότητας ε, παροπλισμού και του ποιο ποσοστό σκαφών αντιπροσωπεύουν κτλ. Είναι απίθανο λοιπόν, αλλά υπάρχει κίνδυνος, αλλά και αν ε, ισχύσει κάτι τέτοιο, θα μπορούσαμε να κάνουμε τον κανονισμό μας να τεθεί σε ισχύ νωρίτερα. Αν προκύψει το σενάριο που επαναλαμβάνω είναι μάλλον απίθανο. Άρα νομίζω ότι είναι ασφαλές να προτείνουμε την επικύρωση αυτής της σύμβασης για σε παγκόσμιο επίπεδο ακόμη και αν τα πρότυπα της ε, σύμβασης του δεν είναι αρκετά για το ευρωπαϊκό επίπεδο και χρησιμοποιούμε αυτή τη σύμβαση ε, για να κάνουμε πιο αυστηρά τα πρότυπα, γιατί επιτρέπεται, κάποια χώρα μπορεί να πάει πιο πάνω από αυτά τα πρότυπα, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο σίγουρα η βελτίωση είναι σημαντική από πολλέ πτυχές, γι' αυτό και συνιστώ να υπερψηφίσουμε την επικύρωση αυτής της σύμβαση. Ο Ευχαριστώ. Δεν έχω τίποτα να πω πέραν της πολύ καλής επεξηγηματικής αιτιολογικής έκθεσης του εισηγητή. Έχει πια ξεπεραστεί από το χρόνο αυτή η σύμβαση, πρέπει να την αναθεωρήσουμε. Βεβαίω είναι καλύτερα από το να μην υπάρχει τίποτα. Βεβαίω όλε αυτέ οι διεθνεί συμβάσει παίρνουν χρόνο για να ε, κυρωθούν. Ε, είναι πολύ βραδύ η χρόνη. Είναι βεβαίω μεγάλη απογοήτευση τη απόρριψη από το κοινοβούλιο τη αρχική πρόταση του Καρλ Σλούτερ. Και βεβαίω υποστηρίζω τα όσα είπε και τι συστάσει του. Σας ευχαριστώ η Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Σλίτσερ ε, περιέγραψε πολύ σωστά στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Έχουμε αυτό τον κανονισμό με βάση την ανακύκλωση των πλοίων που εφαρμόζεται όμως μόνο σε πλοία με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ το θέμα το έχουμε προσυζήτηση διότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρον και σοβαρό και σημαντικό είναι να αναπτυχθεί και η διεθνής ευθύνη, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει αυτή η σύμβαση του Χονγκ Κόνγκ. Υπάρχουν διάφορες πτυχές που πρέπει να υπογραμμίσουμε, δύο κυρίως, ότι μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την ανακύκλωση των πλοίων και για το θαλάσσιο περιβάλλον βεβαίω. και η ε, δεύτερη επίπτωση είναι ότι εξασφαλίζεται ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού για να έχουμε και ένα καλό σύστημα ανακύκλωσης, καλό για το περιβάλλον. Εμείς λοιπόν υπενθυμίζουμε ότι έχει ζητήσει η Επιτροπή την υποχρεωτική προσχώρηση στη σύμβαση και στους όρους της σύμβασης για τα κράτη-μέλη, το οποίο δεν δέχτηκαν όλα τα κράτη-μέλη, έγιναν μακροσκλήσεις στο Συμβούλιο. Πάντως τώρα έχουμε καλή εξέλιξη. Είναι διτεθειμένα τα κράτη-μέλη να ανακυρώσουν αυτή τη σύμβαση και εσείς κύριε Σλίτερ βλέπετε ότι έχει προχωρήσει αυτή η πρόταση. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε στο δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα και ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία πριν από το τέλος της φοιτείας, ε, διότι κράτη-μέλη που περιμένουν την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας υπάρχουν, περιμένουν δηλαδή να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να ξεκινήσουν τη διαδικασία της κύρωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται τη συζήτηση και για αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Στις 4 το απόγευμα σήμερα έχουμε την πρόθεση σημεία για την κατάθεση των τροπολογιών. 16 ε, Μαρτίου ψηφοφορία, 12, ε, και μετά 12 Μαρτίου για την Ολομέλεια κατά πάσα πιθανότητα και μετά έχω την προφορική ερώτηση από το Χάση για το πρόγραμμα βελτίωση τη καταλληλότητα και τη αποδοτικότητα του κανονιστικού πλαισίου, REFIT τη Γενική Νομοθεσία για τα τρόφιμα και το ρόλο του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την καλύτερη λειτουργία τη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Προφορική ερώτηση, όπω είπα. Κύριε Πούλε, όχι, εσεί. Κύριε Σμίκο. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λάβαμε μια θέση με ερωτήσεων για την πρωτοβουλία Refit σε σχέση με το Γενικό Δίκαιο τροφίμων Και βέβαια, αφού κάνω την παρουσίασή μου, μπορείτε να μου θέσετε ερωτήματα για διευκρινήσει. Γνωρίζετε ότι αυτή η πρωτοβουλία κατά βάση εξετάζει τη λειτουργία του υφιστάμενου νομικού πλαισίου από το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων. Πολλοί νόμοι εγκρίθηκαν, πολλά νομοθετήματα ε, εδώ και κάποιο καιρό και θέλουμε να δούμε κατά πόσον πλέον είναι προσαρμοσμένο το νομικό πλαίσιο για τον στόχο που ήθελε να υπηρετήσει. Η γενική λοιπόν λογική της πρωτοβουλίας REFIT είναι αυτή. Στον τομέα των τροφίμων, όπως γνωρίζετε, είναι πολύπλοκο το νομικό πλαίσιο Έχουμε πολλά νομοθετικά πρότυπα αλληλοσυνδεόμενα μεταξύ τους. Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε την πρώτη φάση, fitness first check phase. Δημοσιοποιήσαμε ένα έγγραφο το Δεκέμβριο που περιγράφει το γενικό πλαίσιο και τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σε αυτή την άσκηση REFIT. Και ξεκάθαρα καταδείχθηκε ότι δεν θα είχε νόημα να επικεντρωθούμε σε ατομικά πρότυπα και κανόνες ε, αλλά από τη βάση που διέπει το Γενικό Δίκαιο περί Και στη Γενική Γραμματεία το έχουμε πει ότι ο στόχος μας είναι το γενικό δίκαιο περιτροφίμων, γενική νομοθεσία Περιτροφήμων. Εσείς όμως ε, ρωτάτε λεπτομέρειες. Ε, πρέπει να σας πω ότι ακόμη είμαστε στην προπαρασκευαστική φάση αυτού του εγχειρήματο. Ε, θα προβούμε σε δύο εξωτερικές αξιολογήσεις. Ε, η μία για τον κανονισμό 178 του 2002 και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές είναι το δεύτερο. Ξέρετε ότι υπήρξαν πολλά σκάνδαλα, απάτες με τρόφιμα και πρέπει να δούμε αν ε, στο πλαίσιο αυτού του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα που προέκυψαν με τις τελευταίες αυτές εξελίξεις. Φυσικά και γνωρίζουμε ότι σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να έχουμε και μία ανατροφοδότηση, ένα feedback από τους ενδιαφερομένους. Έξω και η διαδικασία ε, από την αρχή είναι πάρα πολύ διαφανή, συμμετέχουν όλοι γιατί θέλουμε να συμμετέχουν και όλα τα κράτη-μέλη, εμπειρογνώμης από τα κράτη-μέλη, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι, ενδιαφερόμενοι φορείς, είτε φορείς εκμετάλλευσης είναι αυτοί, είτε καταναλωτές, απλοί πολίτες, ΜΚΟ κτλ. Εξού και ήδη ξεκινήσαμε τη διαδικασία, συνεδριάσαμε με τα κράτη-μέλη στις 3 Μαρτίου, ήταν αυτή η συνεδρίαση και θέλω να τονίσω κάτι ακόμη. Πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ χρήσιμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει από την αρχή σε αυτή τη διαδικασία. Καλέσαμε λοιπόν, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρωτοβουλία αυτή, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε, τουλάχιστον μέχρι τώρα, καμία συμμετοχή, ισχύει όμως πρόσκλησή μας ακόμη. Θα διαβολευτούμε λοιπόν με τους εμπλεκομένους ε, στο πλαίσιο της γνωμοδατικής ομάδας, συμπλευτικής ομάδας για την υγεία ε, φυτών ζώων και Γι' αυτό είπα ότι είναι σημαντικό. Έχουμε 45 συμμετέχοντε στην ε, συμβουλευτική αυτή ομάδα. Είναι περιορισμένη σύνθεση, αλλά η ομάδα ε, του Refit είναι ανοιχτή για όλου, ακόμη και όσο δεν είναι μέλη τη συμβουλευτική αυτή ομάδα. Γι' αυτό σα είπα ότι θέλουμε να συμμετέχετε κι εσεί. Στο πλαίσιο αυτή τη συζήτηση ε, προέκυψαν κάποιες προτάσεις για τα στοιχεία της γενικής περιτροφήμων νομοθεσίας που θα πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας. Και αυτά τώρα τα σημαίνει συζήτηση με όλους τους ενδιαφερομένους φορείς. Οι συζητήσει αυτές θα ολοκληρωθούν στις 14 Μαρτίου και βάσει αυτών θα καταλήξουμε στα ζητήματα που θα αξιολογηθούν και θα συνεχίσουμε με εξωτερικές μελέτες που θα διενεργήσουμε το Μάιο. Και ελπίζουμε το 14 περί τα τέλη του έτους να έχουμε τα αποτελέσματα. Έπειτα θα έχουμε τη συνέχεια, ένα follow-up, αλλά αυτό θα βασιστεί και στα πορίσματα, στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων. Άρα προς το παρόν δεν έχουμε προχωρήσει σε κάποια νομοθετική αναθεώρηση, αλλά ε, πρόκειται για μια άσκηση αξιολόγησης που θα μας δείξει σε ποιο επίπεδο η Γενική Περιτροφή Μονομοθεσία ε, μπορεί να εκπληρώσει το στόχο της. Και μόνο ε, ε, μετά από αυτό θα δούμε αν χρειάζεται να, έχουμε, να προβούμε σε περαιτέρω ε, διαδικασίες, να ακολουθήσουμε και άλλα βήματα. Αυτά και είμαι διαθέσιμος να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ο Κάρς Ρούτερ θέλει το λόγο. Ε, ναι, είπαμε, είναι η μέρα μου. Η Σάτου χάσει, έχει υποβάλει αυτή την προφορική ερώτηση, αλλά μου ζήτησαν να την εκπροσωπήσω σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την απάντησή σας. Οι ανησυχίες που είναι και λόγος για την κατάθεση αυτής της προφορικής ερώτησης είναι σαφής. Φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούν με την ανάγκη Προσωπικά, αν ε, θέλω να γελάσει το ακροατήριό μου, διαβάζω τα ποιότητα, ποιοτικά πρότυπα για τα ασπεριδοειδή. Από τα λίγα που παραμένουν στον με των τροφίμων. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή σε αυτό το φόρουμ ψηλού επίπεδου, οι μεγάλες εταιρείες ε, συμμετέχουν. Ενώ εσείς λέτε ότι το 9% είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο. Άρα και περισσότερες ε, επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες. Ερωτώ λοιπόν, υπάρχει ισορροπία ΜΚΟ, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή μεγάλες επιχειρήσεις σε αυτό το φόρουμ. Και είπατε ότι είναι ανοιχτή η πρόσκληση προς όλου αλλά ένας γείτονα που έχει ένα μικροσφαγείο θα έρθει σε αυτό το φόρουμ και μπορεί ακόμη, έχει χρόνο, ε, έχει χρήματα. Οι πολύ μικρέ επιχειρήσει είναι τόσο οργανωμένε ώστε να μπορούν να στείλουν κάποιο σε αυτό το φόρουμ, να πληρώσουν και κάτι τέτοιο. Άρα και πάλι μπορεί να υπάρχει μη ισομερή εκπροσώπηση όλων των ε, εμπλεκομένων στον κλάδο. Και ποιο είναι το βασικό πλεονέκτημα για τις μικρότερες επιχειρήσεις να υπάρχει λιγότερο βάρος, λιγότερο φόρτος. Ο τον μου δεν μπορεί να εξαγάγει ε, το, τα προϊόντα του εκτός ε, της χώρας, μόνο σε τοπικό επίπεδο δραστηριοποιείται. Πρέπει επίσης να πω ότι η εθνική ερμηνεία ορισμένων νομοθετημάτων πολλές φορές δημιουργεί ένα τεράστιο φόρτο για τις ε, μικρές επιχειρήσεις που ε, πολλούν σε τοπικό επίπεδο. Και επειδή δεν υπάρχει διάσταση ευρωπαϊκή ή εθνική, πιστεύω ότι θα έπρεπε οι τοπικές αρχές εδώ να έχουν λόγο. Άρα, επαναλαμβάνω, το όφελος θα το έχουν πιο πολύ οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες ε, και λόμπι ασκούν και μπορούν να προσαρμοστούν πιο εύκολα. Άρα, με ανησυχεί αυτή η έλλειψη ισορροπίας, αν βέβαια υπάρχει τέτοιο πρόβλημα και αν μπορούν να επηρεάσουν και η ΜΚΟ λοιπά. Και είπατε ε, ότι καλείται κάποιε εταιρισμοί, πως καλούνται συγκεκριμένες εταιρείε ή υπάρχει μια γενική εκπροσώπηση των μεγαλύτερων εταιρείων. Δεύτερη μέρημνά μας είναι υπάρχουν αρκετές εγγύησεις ώστε να μην είσαι αρχή της προφύλαξης. Και η μείωση των βαρών να είναι μείωση των βαρών και όχι μείωση στον τομέα της ασφάλειας ή της περιβαλλοντικής προστασίας. Η Επίτροπη παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα πρέπει καταρχά να πω ότι αντιλαμβανόμαστε την γνώση αυτών των ανησυχών και τις παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει σημαντική, σημαντικό ποσοστό μικρών επιχειρήσεων στον χώρο των τροφίμων, στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα παρακολουθούμε ε, την δυνατότητα προσώπηση ακριβώς αυτών των επιχειρηματιών. Βεβαίω, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ή να ερμηνευθεί η refit ως περιοριζόμενη μόνο στο φόρουμ υψηλού επίπεδου. Άλλωστε το φόρουμ υψηλού επίπεδου συστήθηκε πριν από μερικά χρόνια από τους συναδέλφους Γενικής Διεύθυνσης ε, για τις επιχειρήσεις για άλλο θέμα, σε άλλο τομέα, αλλά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για συνάντηση, για συζήτηση με τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον χώρο των τροφίμων και πράγματι και εμείς αυτή την πρόκληση την αναλαμβάνουμε. Χρησιμοποιούμε αυτό το φόρουμ, αυτό το κέντρο συζητήσεων για ανταλλαγές απόψεων σχετικές με συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες, νέες νομοθετικές προτάσεις και αυτό όχι μόνο για τη συγκεκριμένη ρέφητα, αλλά διαρκώς. Άρα έχουμε αυτή τη δυνατότητα, το φόρουμ υψηλού επίπεδου, που αξιοποιούμε, που δεν είναι όμως και ο μόνος εταίρος στο εγχείρημα αυτό που ονομάζεται Refit. Έχουμε μια ομάδα συμβουλευτική, όπου η εκπροσωπήση τόσο καταναλωτών όσο και μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι πολύ ψηλή. Άνω του ίμιση των συμμετεχόντων, αν δεν απατώμε, σε σχέση με παρουσία φορέων και όπως είπα έχουμε συστήσει αυτή την ομάδα εργασίας στην οποία είναι ανοιχτή η πρόσβαση για τους πάντες. Ε, βέβαια το θέμα είναι πώς μπορεί ένας ε, παράγων από μικρή επιχείρηση να μπορέσει να ενταχθεί σε αυτή τη διαδικασία. Εκείνη η δυσκολία και συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε την εκπροσώπηση από τους καταναλωτές, οι οργανώσεις των καταναλωτών. Πολύ συχνά με τις τοποθετήσεις τους εγείρουν ζητήματα συμφερόντων των μικρότερων επιχειρήσεων. Και έχουν, οφείλω να πω, τη δυνατότητα οι εκπροσωπήσεις, οι εκπρόσωποι των καταναλωτών έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπηση. Έχουν περισσότερου δηλαδή εκπροσώπους από η άλλη ομάδα συμφερόντων. Πέραν αυτού, έχουμε και την πρόθεση για πιο στενή συνεργασία, γιατί είναι πολλά και τα κράτη-μέλη που ενδιαφέρονται για αυτή την ε, πρωτοβουλία και που θα μπορούσαν ε, να λάβουν μέρος σε πιο λεπτομερείς αναλύσεις σε διαφορούς τομείς. Όπως γνωρίζετε, παραδείγματι, το έχουμε ήδη δει και στις κατοχώρες, στον χώρο των ε, αρτο, της αρτοποιίας, όπως άλλωστε θα το δούμε και στο Ηνωμένο Βασίλειο σύντομα και πολλές άλλες πληροφορίες μπορούν να ενταχθούν σε αυτή την πρωτοβουλία. Για την ερώτηση σας τώρα για την ε, ε, αμφισβήτηση ημί των βασικών αρχών. Δεν είναι αυτό ζήτημα του Ρέφιτ. Η πρόθεση δηλαδή, του Ρέφιτ δεν είναι να αμφισβητήσει τις αρχές, αλλά να εξετάσει εάν οι πρακτικές που υπάρχουν εξυπηρετούν τους αρχικούς στόχους, όπως είχαν οριστεί, τις αρχικές προθέσεις. Δηλαδή, η νομοθεσία όπως έχει σχεδιαστεί, όπως είχε σχεδιαστεί το 2002, εξυπηρετεί ακόμη τους στόχους εν έτη 2014, όπως αρχικά είχε προβλεφθεί. Και αυτό γιατί έχουν ε, μεταξύ παρασφρήσει εξελίξεις, νέα στοιχεία, υπάρχουν παρατηρήσεις. Αυτό λοιπόν. Και σας διαβεβαιώ ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να μειώσουμε το επίπεδο της ασφάλειας των τροφίμων, της ασφάλειας που αισθάνεται ο καταναλωτής στον τομέα αυτόν. Αλλά αποδεχόμαστε και το γεγονός ότι κάποιες εξελίξεις μπορεί να αλλάξουν τις συνθήκες και άρα μπορεί να αναζητήσουμε έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο για την υλοποίηση αυτής της ε, αντίληψης περί ασφάλειας. Και βεβαίως άπαξ και δούμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, άπαξ και αντιληφθούμε πώς ε, γίνεται αντιληπτή από την πρακτική έποψη τα κράτη-μέλη, τους διαφορούς φόρους κτλ. η νέα νομοθεσία για τα τρόφιμα, τότε μόνο μπορούμε να ορίσουμε εάν διότι μπορεί να προκύψει αποτέλεσμα είτε ότι όλα πάνε καλά ή ότι όλα πάνε όσο καλά θα μπορούσαν να πηγαίνουν και άρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα ή δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα. Είναι πολύ πιθανό να προκύψει αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ δεν είμαι σε θέση να προβλέψω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής. Θα δούμε στα τέλη του 2014. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Εξαντληθήκε η μυρίσια διάταξη. 10 Μαρτίου. Προσεχή. Τρίτη δηλαδή, έχουμε την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας στο Στρασβούργο. από τις 6 μέχρι τις 10.30 με πολύ πλούσιο πρόγραμμα, καθόλου βαρετό. Θα έχουμε προσκεκλημένους 19 Μαρτίου 9 μέχρι το 12.30 3 με 6.30, 14 Απριλίου τελευταία συνεδρία της Επιτροπής από τις 7 έως τις 10.30 και ολοκληρώνεται έτσι η θητή αυτή. Τελειώνουμε λοιπόν προς το παρόν τη Δευτέρα. Θα τα πούμε και ευχαριστώ όλους τους παρισταμένους.